Dear colleagues, dear friends, please take your seats and, and let's get started. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Έχουμε αργήσει ήδη λίγο. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο, μόνο δεν είχαμε χρόνο στις 27 Ιουνίου, οπότε με γραπτή διαδικασία πήραν κάποιες αποφάσεις οι συντονιστές όσον αφορά τις Ισπανικές Τράπεζες με ψήφισμα. Το ΕΛΚ ζήτησε να ψηφιστεί η απόφαση των συντονιστών, οπότε θα επανέλθουμε σε αυτό. Σε λίγα λεπτά. Δεύτερον, τη από τις ομάδες. Υπάρχει για την 1555 Παύλα 12 ένα αίτημα όπου οι συντονιστές αποφάσισαν να προωθήσουν αυτή την αναφορά στην Εύη και Ήτρε και θα το συζητήσουμε όταν λάβουμε τις γνωμοδοτήσεις Εύη και Ήτρε. Επίσης για την 0098 Παύλα 15 κατεπήγουσα διαδικασία και αποφασίσαμε να την συμπεριλάβουμε στην ε, διαδικασία της ε, συνεδρίασης μας το Σεπτέμβριο μαζί με άλλα θέματα αναπηρίας. 0112 Παύλα 15 αποφασίσαμε να την αντιμετωπίσουμε μαζί με άλλες εκκρεμούσες αναφορές τον Οκτώβριο ή αργότερα εντός του 15 κατόπιν για την 2158 Παύλα 14 αποφασίσαμε να μπει στην ημερήσια διάταξη του Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε θα έχουμε και την ενημέρωση ελπίζουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπουμε επίσης συμφωνήσαμε να ζητήσουμε το Τμήμα Πολιτικής να μας κάνει μια μελέτη για τις αναπηρίες. Κατόπιν είχαμε προφορική και γραπτή ενημέρωση για τη δικτυακή πύλη της ΠΕΤΗ και ζητήσαμε, αποφασίσαμε να ζητήσουμε από την νομική υπηρεσία να μας διευκρινίσει ορισμένα θέματα ιδιωτικής σφαίρας και ε, προστασία δεδομένων για το άνοιγμά της σε όλα τα μέλη. Επίσης, τα αιτήματά μας για το πρόγραμμα εργασίας του Ελεκτικού Συνεδρίου. Αποφασίσαμε ότι τα αιτήματα των ε, ομάδων θα αποσταλούν στο πρόγραμμα εργασίας του Ελεκτικού Συνεδρίου και ο διαφρομένος διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία συνοπτική έκθεση και εκκλήσεις για δράση. Θα στείλουμε πέντε προτεραιότητες για να μπουν στο πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2016. Θα τα στείλουμε αυτά μέσω τη διάσκεψης των Προέδρων, των Επιτροπών. Κατόπιν, έχουμε σήμερα το πρωί λάβει μία απόφαση ως συντονιστές. Πρώτα απ' όλα εγκρίναμε την ε, ημερήσια διάταξη για τη συνεδρία της 17 Σεπτεμβρίου με κάποιες τροποποιήσεις. Το σημείο 8, η έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΠΕΤΗ, αποσύρθηκε. Θα επανέλθω μετά γι' αυτό. Και το 10 που είναι η 0481 του 13 αναφορά επίσης αφαιρέθηκε και αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο διότι η Επιτροπή δεν ήταν έτοιμη να μας υποβάλει πλήρη ενημέρωση το Σεπτέμβριο αλλά θα μας την έχει αποστείλει πριν την συνεδρίασή μας του Οκτωβρίου. Επίσης συντονιστές συμφώνησαν ότι σε επόμενες ημερήσεις διατάξεις θα συμπεριληφθούν τα εξής. τον Οκτώβριο η 0884 του 14 και τον Νοέμβριο η 1156 του 13 και η γνωμοδότηση για την έκθεση για τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγγνώμη τη Σύμβαση των Ηνωμένων για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αποφασίστηκε να υπάρξει μια γνωμοδότηση τέσσερα για το θέμα αυτό μαζί με την ΛΥΜΠΕ, την Επιτροπή, όχι λάθος, όχι ΛΥΜΠΕ, την Επιτροπή Απασχόλησης και η Ρώσα Εσταράς Φεραγκού του ΕΛΚ θα είναι η συντάκτρια. Και επιβεβαίωση ότι η συγητής για την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του διαμεσολαβητή θα είναι η Σολεδάδ Cabezón Ρουίθ και δεν θα υπάρξει νομοδότηση με βάση το άρθρο 54 για το γενικό προϋπολογισμό γιατί μόνο μία γραμμή του προϋπολογισμού μας αφορά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης εγκρίναμε το αίτημα για μια σύντομη μελέτη από το Τμήμα Πολιτικής για τα θέματα που θέτει η αναφορά για την ενεργειακή πολιτική μέσω ηλιακής ενέργειας στην Ένωση και τα κράτη-μέλη. Και επειδή υπάρχουν διαφωνίες επί των συστάσεων, το αναβάλαμε για το Σεπτέμβριο. Η συνέχιση της ενασχόλησής μας με το Jugendamt και αποφασίσαμε γι' αυτό να δημιουργηθεί ένα μια ομάδα εργασία. Το Jugendamt είναι η Υπηρεσία Προστασία Ανηλίκων τη Ομοσπονδιακή Γερμανία. Και θα διευρύνουμε το πεδίο ενδιαφέροντο σε γενικότερα θέματα ευημερία των παιδιών με βάση τις αναφορές που έχουμε λάβει. Επίσης, θα ασχοληθούμε με άλλα θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά. Για παράδειγμα, αυτό το Jugendamt, διεθνεί απαγωγέ παιδιών, δηλαδή από χώρα σε χώρα, υποχρεωτικές υιοθεσίε κτλ. Σε αυτή την ομάδα εργασίας θα συμμετάσχει ένα μέλος αναπολιτική ομάδα και ανεξάρτητα θα αποφασίζει για τις μεθόδους εργασίας της και θα καθορίζει τον πρόεδρο της ομάδα εργασίας. Και τα απορίσματα πρέπει να μας υποβληθούν πριν από την δεύτερη του Σεπτεμβρίου. Συγγνώμη, πριν, ναι, τη 2 Σεπτεμβρίου. Επίσης, αποφασίσαμε ότι στη δικτυακή μας πύλη θα μπαίνουν τα πρακτικά και το web streaming και, θα, και επιβεβαιώθηκε το σύστημα που έχουμε για την συνυπογραφή αναφορών. Επίσης πήραμε μία απόφαση να κάνουμε τρεις διερευνητικές επισκέψεις το δεύτερο εξάμεινο του 2015 και το πρώτο του 2016. Πρώτη στον νόμιμο Βασίλειο. 3 με 6 Νοεμβρίου στην Ισπανία, στη Μαδρίτη συγκεκριμένα, την περιοχή των, των ποταμών Εύρο και Τάχο 8 με 12 Φεβρουαρίου και ε, επίσης στην Ιρλανδία την άνοιξη του επομένου έτους ως γενικό κανόνα. Επίσης αποφασίσαμε ότι για κάθε τέτοια αποστολή θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τέσσερα μέλη. Αλλά η αποστολή μας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πολύ πιο διευρυμένη. Μπορούν να συμμετάσχουν 12 μέλη και τα ονόματα των ενδιαφερομένων πρέπει να μας αποσταλούν πριν τις 15 Σεπτεμβρίου. Ακρόαση τώρα για τις αναπηρίες. Εγκρίναμε το πρόγραμμα. Θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου το πρωί αυτή η ακρόαση. Μας ενημέρωσε η νομική υπηρεσία για την αναφορά 570 Παύλα 13 η, γενική υπηρεσία, η νομική υπηρεσία συγγνώμη, μας παρουσίασε τις ε, νομικές επιλογές με βάση τον κανονισμό, την ομολογία και τις συνθήκες. Και οι συντονιστές ε, επιφόρτησαν τη γραμματεία να εξετάσει την συνέχιση που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτήν την αναφορά. Και στα διάφορα ο κύριος Μαριάς μας παρουσίασε μία νέα επιγραμμική πλατφόρμα την οποία κατήρτισε και για ενημέρωση. Έχει το κατάλογο 3 για το ποιες αναφορές θα μπορούσαν να θεωρηθούν απαράδεκτες το ε, χρονοδιάγραμμα για τις εκθέσεις για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και το ε, χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεών μας. Και κατόπιν είχαμε μία μακροσκελή ανταλλαγή απόψεων για τις ε, υποεξέταση κατευθυντήριες γραμμές. Σημειώσαμε ότι δύο τεχνικές συνεδριάσεις έχουν ήδη διεξαχθεί για να υπάρξει ένα αναθεωρημένο κείμενο ως βάση συζήτησης. Αυτή η αναθεωρημένη βάση θα υποβληθεί το Σεπτέμβριο στους συντονιστές και στην Επιτροπή μας, ελπίζω για έγκριση, ήδη τον Οκτώβριο. Αυτά συζητήσαμε το πρωί. Και τώρα, επειδή το 6 αναβλήθηκε για το απόγευμα, να ψηφίσουμε την απόφαση των συντονιστών να υποβληθεί ψήφισμα σχετικά με την Ισπανική νομοθεσία για τι υποθήκε και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου. Έχει ζητήσει το ΕΛΚ να ψηφίσουμε όλη την απόφαση των συντονιστών να εγκρίνουμε ψήφισμα ω Επιτροπή. Μία ψηφοφορία λοιπόν θα γίνει. Ελπίζω να έχετε τις κάρτες σας, γιατί μπορεί να χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουμε. Αλλά ίσως για αυτήν την ε, ψηφοφορία ε, να μην χρειαστούν. Να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Υπέρ λοιπόν του να συνταχθεί αυτό, αυτή η πρόταση ψηφίσματος. Παρακαλώ, σήκωστε τα χέρια σας. Κατά Αποχές. Μία αποχή. Ωραία. Ευρία πλειοψηφία λοιπόν. Και μία ομάδα βέβαια είναι εντελώς αντίθετη. Αλλά όπως κάθε δημοκρατικό σώμα έχει εγκριθεί η απόφαση αυτή. Δεύτερη ψηφοφορία που νομίζω ότι πρέπει να είναι ηλεκτρονική είναι η προφορική ερώτηση για αυτά τα θέματα στην Ισπανία, υποθήκες και χρηματοπιστωτικά προϊόντα ψηλού κινδύνου. Έχει συμφωνηθεί ένα συμβαστικό κείμενο ε, S&D, άλτεγκου και Πράσινη. Έχουμε εδώ το κατάλογο ψηφοφοριών. Πρώτον, συμβαστική τροπολογία Α. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά συμβαστική τροπολογία Β, S&D, Αλτεγκού και Πράσινη. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και έτσι λίγη Δεν υπάρχει άλλη τελική ψηφοφορία. Έτσι λίγη ψηφοφορία. Όχι. Δεν βλέπω εδώ στον κατάλογο ψηφοφοριών. Πρέπει στο τέλος να υπάρξει τελική ψηφοφορία. Πρόεδρος, λέω, εφόσον υπάρχει ψήφισμα ή νομοθέτημα πρέπει να υπάρξει τελική ψηφοφορία. Αλλά αυτό είναι προφορική ερώτηση. Δεν χρειαζόμαστε τελική ψηφοφορία. Υπάρχει τώρα το τροποποιηθέν και εγκριθέν κείμενο. Νομίζω ότι με βάση οποιαδήποτε διαδικασία έχουμε αξιοποιήσει μέχρι τώρα, αυτό κάνουμε. Αλλά ο Πέτερ έχει το λόγο. Μία παράκληση και μία παρατήρηση. Η παράκληση στο μέλλον όταν θέλουμε να τροποποιήσουμε την ημερήσια διάταξη να μην γίνεται με γραπτή διαδικασία είναι μέτρο έκτακτης κατάστασης το κάναμε αλλά παρακαλώ στο μέλλον ε, να μην γίνονται τέτοια πράγματα να το συζητάμε είτε ως Επιτροπή είτε ως συντονιστές και επίσης θέλω να πω ότι λυπάμαι ιδιαίτερα που δεν ε, συμπεριλήφθησαν στην ε, συμβαστική πρόταση B η προτάσει τη ομάδας μου, γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να απορρίψουμε τη συμβαστική τροπολογία B. B. Πρόεδρος. Μα έχετε κάθε δικαίωμα. Κάθε δικαίωμα να καταψηφίσετε, αλλά παρόλα αυτά εγκρίθηκε. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι χρειάστηκε να υπάρξει γραπτή διαδικασία γιατί προβλέπουμε πολύ λίγο χρόνο για τους συντονιστές σε σχέση με άλλες επιτροπές. Στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε ένα πιο λογικό χρονικό διάστημα για τους συντονιστές γιατί όλο και περισσότερες αποφάσεις πάνε στους συντονιστές. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για όλους τους συναδέλφους συντονιστές Οπότε μέσω της Βύρπη εδώ και της γραμματείας ε, συνολικότερα θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε περισσότερο χρόνο για τους συντονιστές από το φθινόπωρο. Άψογα. Η Σολεδά. Πολύ σύντομα θέλω να διευκρινίσω κάτι. Καταλαβαίνω την ε, θέση του ΕΛΚ αλλά νομίζω ότι όλοι προσπαθήσαμε να συμφωνήσουμε και να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Εκατό λέξεις μπορούσαμε να βάλουμε μόνο στο κείμενο, ήμασταν περιορισμένοι, οπότε δεν μπορώ να δεχτώ ότι τίποτα δεν συμπεριλάβαμε, γιατί η τελευταία ερώτηση είναι ακριβώς αυτό που ζήτησε το ΕΛΚ. Υπήρξε πολύ καλή βούληση, αλλά οι περιορισμοί είναι περιορισμοί στο κείμενο. Τίποτα άλλο, αυτό μόνο ήθελα να πω. Άλλος κανείς που θέλει το λόγο από αυτού. Παρακαλώ. Ρώσα. Δεν συμφωνώ με τα τελευταία που ακούσαμε από την φίλη Σολεδάτ. Νομίζω ότι στην πράξη τίποτα δεν ε, δεχτήκαμε από αυτά που ζητήσαμε. Άλλαξε επίση η ημερήσια διάταξη επειδή ένα βουλευτή από κάποια ομάδα έστειλε κάτι γραπτά ή όχι. Έχουμε περάσει όλο το πρωί το απόγευμα πάνω σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα στο μέλλον να το συζητάμε, να ξέρουμε πότε θα ψηφίσουμε ακριβώς πρωί απόγευμα και οι προτάσεις του ΕΛΚ δεν έγιναν αποδεκτές. Είμαστε κατά και εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολιτική πρωτοβουλία ουσιαστικά και που δεν εξυπηρετεί τους πολίτες. Ευχαριστώ. <coughs> Πρόεδρος, άλλος. Ωραία. Θέλω να υπογραμμίσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 128 του κανονισμού είναι η διάσκεψη των Προέδρων που αποφασίζει πότε και με ποια σειρά ε, μπαίνουν ε, τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Οι ερωτήσεις που σε τρεις μήνες δεν έχουν μπει στην ημερήσια διάταξη ε, φεύγουν. Πριν από την σύνοδο ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για το με ποια σειρά θα υποβληθούν. Είχαμε διάφορες συζητήσεις μέχρι τώρα για τα διάφορα θέματα. Μερικές φορές πρέπει απλώς να κοιτάμε κατάματα την πραγματικότητα. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Δεν συμφωνούν όλοι πάντα, ούτε έχουμε όλοι πάντα την ίδια θέση. Αυτή είναι η πολιτική και μερικές φορές πρέπει απλώς να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Η πλειοψηφία τώρα πήρε την απόφαση που πήρε. Οπότε, τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε το ψήφισμα για τις υποθήκες χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου στην Ισπανία και να συντάξουμε ψήφισμα. Λοιπόν, έχετε το κείμενο μπροστά σας. Οπότε, ποιος θέλει το λόγο. Επί του κειμένου αυτού. Σολεδάδ. Ευχαριστώ. Ένα τεχνικό ζήτημα. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι μέχρι την επόμενη εβδομάδα στις 21 του μηνός. Είναι δυνατόν να παρατείνουμε λίγο αυτή την προθεσμία. Ωραία, έχει ως εξής το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών ήταν πράγματι αρχικά 20 Ιουλίου. Άλλαξε, έγινε 24 Ιουλίου τώρα. Η έγκριση θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου, τότε θα ψηφίσουμε και κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο ή και αργότερα θα περάσει από την Ολομέλεια. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Συνεπώς, αυτό που έχετε μπροστά σας τώρα είναι το κείμενο το οποίο έχει ετοιμάσει η Γραμματεία. Και είσαστε ελεύθεροι, μπορείτε κάλλιστα μέχρι τις 24 Ιουλίου να υποβάλλετε τροπολογίες από αυτού. Εντάξει, Πίτερ. Παρακαλώ τους συναδέλφους ε, να με καταλάβουν. Και εγώ πάντα λέω ότι η προφορική ερώτηση χωρίς ψήφισμα δεν έχει έννοια. Όμως, η ομάδα μου αυτή τη φορά προτείνει πρώτα να συζητηθεί στην Ολομέλεια η προφορική ερώτηση και κατόπιν μαζί με τις άλλες καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές να επιχειρήσουμε να συντάξουμε ψήφισμα γιατί ξέρετε υπάρχει κίνδυνος να γίνει πολύ έντονη συζήτηση Και μπορούμε βέβαια να κρίνουμε και ψήφισμα και μετά όλα να ηρεμήσουν. Αλλά αν θέλουμε κάτι να αλλάξουμε ως Επιτροπή Αναφορών, τότε πρέπει να συνεργαστούμε με τις άλλες ομάδες. Γι' αυτό είχαμε πει ως ομάδα πρώτον η συζήτηση της προφορικής ερώτησης και μετά να δούμε με τις ε, αρμόδιες επιτροπές να δούμε εάν έχει ένα να υπάρξει ψήφισμα. Μόνο έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση. Σας το λέω παρόλο που σας λέω ότι γενικά η άποψή μου ε, είναι διαφορετική από αυτό το θέμα. Μίσες Βαλίνα. Η κυρία Βαλίνα. Όπως είπε και η Σολεδάδ και εγώ το ίδιο ήθελα περισσότερο χρόνο για τις τροπολογίες το Σεπτέμβριο τουλάχιστον γιατί 17 με 24 είναι σύντομο το χρονικό διάστημα αν γίνεται να παρατείνουμε λίγο παραπάνω την προθεσμία. Η κυρία Αλμπιόν. Ευχαριστώ. Θέλω να υπογραμμίσω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό να πάει στην Ολομέλεια και να υπάρξει ψήφισμα από την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου το ψήφισμα να αντικατοπτρίζει αυτό το οποίο καταγγέλουν ακριβώς οι αναφέροντες. Υπάρχουν 20 για τις υποθήκες και καμία για τα προτιμησιακά. Συνεπώς, το ψήφισμα πρέπει να αντικατοπτρίζει ακριβώς το δράμα που έχουν ζήσει τόσοι πολίτες στην Ισπανία τα τελευταία 7 χρόνια, όπου 500.000 υποθήκες χρειάστηκε να πληρωθούν αλλιώς τους σπίτια και θέλουμε επίσης να καταγγείλουμε πώς τα άτομα αυτά τα βγάλαν από τα σπίτια τους επειδή δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να πληρώνουν τις υποθήκες τους, τους έκαναν έξωση και θέλουμε να αναφερθεί και απάτη που έγινε με τις προτιμησιακές εποχές, μετοχές. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις κατάλληλες τροπολογίες για να βελτιωθεί το κείμενο. Ευχαριστώ. Τανόκα, κυρία Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν παρούσα στην ε, ε, προηγούμενη θητεία, 16 Απριλίου, στην Επιτροπή Μεταφορών, ε, συγγνώμη, Αναφορών, όπου συζητήθηκε το θέμα της Ισπανίας. Εν τω μεταξύ όμως άλλαξε ο τίτλος και στα A, ε, θα, στις αιτιολογικές σκέψεις ε, αναφερόμαστε μονάχα στην Ισπανία ή και σε άλλες ε, χώρες γιατί και στη Λετωνία, στη δικιά μου χώρα έχουμε τέτοιου είδους ε, προβλήματα θέλω να το καταλάβω αυτό και βεβαίως και εμείς θα περισσότερο χρόνο για την υποβολή των τροπολογιών όχι, το, το, το, μόνο η Ισπανία αφορά μόνο την Ισπανία το θέμα αυτό σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον we, have voted. Πρόεδρος, ψηφίσαμε πριν από λίγο και επ' αυτού ψηφίσαμε. Αυτό είναι αυτό που βλέπετε, είναι αυτό που ψηφίσαμε. Χωρίς μικρόφωνο. Ναι, αλλά άλλαξε ο τίτλος. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ σαφές ότι αναφερόμαστε στην Ισπανία. Λέγαμε in Spain, ενώ τώρα δεν είναι πολύ προφανές. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά έτσι νομίζω. Πρόεδρος, αν θέλετε να τροποποιήσετε τον ε, τίτλο, έπρεπε να το κάνετε πριν ε, την ψηφοφορία. Όχι, δεν αναφέρουμε μόνο στον τίτλο, αλλά και στις αιτιολογικές σκέψεις. <clears throat> ναι, αλλά τώρα ψηφίσαμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Κύριε Μαριά, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε τρία θέματα. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι συμφωνήσαμε όλοι προηγουμένως και είχαμε μια ψηφοφορία ότι θα έχουμε ψήφισμα. Διότι απλή ερώτηση, προφορική, χωρίς ψήφισμα, σε μια εποχή όπου πραγματικά έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ισπανία, νομίζω ότι θα ήταν λάθος. Επομένως είναι σημαντικό το ότι καταλήξαμε σε απόφαση για ψήφισμα έτσι αν θέλετε στηρίζουμε την προσπάθεια όλων των αναφερόντων που ήρθαν εδώ και έθεσαν το σημαντικό αυτό ζήτημα που υπάρχει στην Ισπανία με τις χιλιάδες εξώσεις και αυτό το τεράστιο κοινωνικό ζήτημα και κυρίως την αυθαιρεσία των διαφόρων τραπεζών. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε το πρώτο θέμα. Δεύτερον, το ψήφισμα έτσι όπως το βλέπω αποτελεί μια σημαντική βάση και νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο να ετοιμάσουμε τροπολογίες για να μπορέσουμε να πάμε όταν θα είναι να συζητηθεί στην Ολομέλεια. Το τρίτο, ε, επιτρέψτε μου ότι ψηφίσαμε βεβαίως τον ε, τίτλο και νομίζω ότι κάναμε δεκτή την τροπολογία που λέει ότι ε, αφορά ε, mortgage legislation and risky financial instruments in the EU, the case of Spain. Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως αφορά την Ισπανία, αλλά στις αιτιολογικές εκθέσεις και στις αιτιολογικές σκέψεις μπροστά, επειδή είναι in the EU, προφανώς και εγώ θα καταθέσω αντίστοιχη τροπολογία, υπάρχουν τέτοια προβλήματα και στην Ελλάδα. Έχουμε προβλήματα με τα στεγαστικά δάνεια, ιδίω με αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, είναι πάνω από 70.000 Έλληνες και αυτοί έχουν προβλήματα. Επομένως, χωρίς να ανατρέπουμε τη φιλοσοφία του ψηφίσματος, στις αιτιολογικές σκέψεις θα το βάλουμε και εμείς από την πλευρά μας και ελπίζω να υπάρχει ανταπόκριση και από τους άλλους συνάδελφους. Το βασικό είναι βέβαια η Ισπανία. Αλλά in the EU στις αιτιολογικές σκέψεις μπορεί να αναφερθεί και η Λετωνία. Νομίζω λοιπόν ότι καταλήγουμε, από εκεί και πέρα έχουμε το χρόνο για τις τροπολογίες, για να συζητήσουμε επιτέλους στην Ολομέλεια, με ψήφισμα, ένα σημαντικό θέμα που υπάρχει σε ένα κράτος μέλος και που ήρθε εδώ μετά από αναφορές από τους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρώστα. Λοιπόν, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα για αυτές τις ε, προνομιακές μετοχές και τι έχουν κοστίσει στους ανθρώπους. Έχει να κάνει και με την Ισπανία και με το τι προστασία υπάρχει για αυτούς που έχουν λάβει ενυπόθηκο δάνειο. Δεν αφορά μόνο την Ισπανία. Αλλά ξέρετε τον Νοέμβριο έχουμε εκλογές στην Ισπανία. Εάν περάσει Οκτώβριο ή Νοέμβριο στην Ολομέλεια και τότε περίπου θα περάσει, τότε θα θεωρηθεί ως πολιτική παρέμβαση στις εκλογές. Γι' αυτό καλύτερα θα ήταν να περάσει σε μια ολομέλεια που να είναι πιο απομακρυσμένη από τις εκλογές. Γιατί αν περάσει τον Νοέμβριο δύσκολα θα μπορέσει να πιστέψει κανείς ότι ε, γίνεται για να προστατεύσει κάποιους και όχι για να παίξει ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία. Πρόεδρος. Όχι, πολλοί θέλουν τον λόγο. Πρώτα η Σολεδάδ. Και μετά πάλι κυρία Βαλίνα. Τώρα για το τεχνικό θέμα και την επιμήκυνση των ε, προθεσμίων θα μπορούσαμε για παράδειγμα να έχουμε προθεσμία μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου για να το εγκρίνουν 17 για να μην καθυστερήσει. Νομίζω ότι κοροϊδεύουμε τους πολίτες εάν τους λέμε ότι δεν κάνουμε πολιτική. Είναι πολιτικά όλα αυτά τα θέματα. Ότι μπορεί να παίξει ρόλο στις πανικές εκλογές. Φυσικά και το αποτέλεσμα για παράδειγμα των ελληνικών εκλογών το Σεπτέμβριο μπορεί να παίξουν ρόλο στις ισπανικές εκλογές. Όλα μπορούν να επηρεάσουν τα πάντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε αυτή τη συζήτηση. Και αν θεωρούμε ότι μπορεί να επηρεάσει τις εκλογές, τότε να φροντίσουμε να μην τις επηρεάσει. Κοιτάξτε, αυτά είχε γίνει τότε και με τους σοσιαλιστές. Αυτά είχαν κάνει οι δεξιοί όταν οι σοσιαλιστές ήταν κυβέρνηση και τώρα είναι η σειρά τους. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να εκφράσουμε τα ανησυχία των πολιτών για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα τους και σε άλλες χώρες βέβαια βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις ε, κακών πρακτικών από τις τράπεζες. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό και πρέπει να βοηθήσουμε να διορθωθούν όλες αυτές οι αδικίες. Γιατί θα χάσουμε τον μπούσουλα. Πρέπει να υπάρξει ψήφισμα, πρέπει να έχουμε στόχους διότι είναι σαφές ότι είναι ανεπαρκής η ισπανική νομοθεσία, δεν έχει μεταγραφεί σωστά η οδηγία 93-13 και αυτό υπάρχει και σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δεν υπάρχει, συγγνώμη, του ανώτατου Ισπανικού Δικαστηρίου και δεν υπάρχει καμία δράση από τις Ισπανικές αρχές για να σταματήσουν, να καταργηθούν δηλαδή αυτές οι καταχρηστικές διατάξεις. Άρα κάτι υπάρχει από πίσω. Είναι αυτό πολύ σημαντικό για την ισπανική κοινωνία, για την ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινωνία και θεωρώ ότι δεν είναι, αδυ... δεν είναι δυνατόν να το αναβάλουμε επειδή επίκυνται εκλογέ. Μα δεν είναι κάτι που μπορεί να βγει από το γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής και των εκλογών. Και νομίζω ότι αυτή η ε, δικαιολογία είναι η χειρότερη πρόφαση για να αναβάλουμε τη συζήτηση. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μπορούμε να μεταφέρουμε αργότερα τον Ιούλιο ή το Σεπτέμβριο την ε, προθεσμία υποβολής των τροπολογιών. Αλλά τότε ε, πραγματικά δεν θα μπορέσουμε να το περάσουμε στην Ολομέλεια κάπου πριν τα Χριστούγεννα γιατί θα πρέπει να μεταφραστούν τα κείμενα κτλ. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να υπογραμμίσω. Δεύτερον, όπως είπα και προηγουμένως, σύμφωνα με τον 128 ε, του εσωτερικού ε, η διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει κατά αποκλειστικότητα ε, τα θέματα τα οποία θα μπουν στην ημερήσια διάταξη. Άρα μην θεωρήσετε κάτι δεδομένο. Ε, εμείς πρέπει να δουλέψουμε απλώς. Η κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι η εντολή που έχουμε από τους πολίτες είναι πολιτική και είμαστε εδώ για να κάνουμε πολιτική. Δεν είμαστε υπάλληλοι, αξιωματούχοι, οπότε υποχρέωσή μας είναι και χρέος μας είναι να υποστηρίξουμε τους πολίτες εκείνους οι οποίοι μας έφεραν εδώ. Είτε υπάρχουν εκλογές τον Νοέμβριο ή τον Ιανουάριο κτλ. Δεν έχει σημασία. Η υποχρέωσή μας είναι αυτό που είναι. Σήμερα το πρωί, Ρώσα, μιλούσες για την πολιτική βούληση για την ταλιδομίδη. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Πρέπει να έχουμε πολιτική βούληση να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Και εξώσεις υπάρχουν κάθε μέρα, χιλιάδες κάθε μέρα. Συνεπώς, οι αναφορές βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό μπροστά μας. Οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα στον κόσμο, είτε υπάρχουν εκλογές είτε δεν υπάρχουν, εμείς να τους υποστηρίξουμε και οι κυβερνήσεις μας, είτε είναι του ΕΛΚ είτε οτιδήποτε άλλο, να τηρούν τις οδηγίες και να τηρούν τον νόμο και να δουλεύουν υπέρ των πολιτών και όχι να βγάζουν στο δρόμο οικογένειες με μικρά παιδιά. Τώρα, αν υπάρχει μια τόσο μεγάλη απάτη όπως είναι εκείνη με τις προνομιακές συμμετοχές, πρέπει να τιμωρηθεί και τα χρήματα πρέπει να επιστρέψουν στους πολίτες. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Τα υπόλοιπα, αν ήμασταν υπάλληλοι, δεν θα ήμασταν εδώ. Εδώ είμαστε για να κάνουμε πολιτική ακριβώς. Πρόεδρος. Και η πολιτική λοιπόν απόφαση που μόλις πήραμε αφορά την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα. Επομένως δεν καταλαβαίνω γιατί ξανασυζητάμε ε, το θέμα. Τώρα θα πρέπει να δεχτούμε ή να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα και μετά να αρχίσουμε να υποβάλουμε τροπολογίες. Τελεία και παύλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχω 7 ε, ε, Ισπανούς που ζητούν το λόγο, ο ένας μετά τον άλλον. Ε, πραγματικά αυτό θέλουμε να κάνουμε ε, σε τούτη την Επιτροπή, ε, μη έχοντας και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Αν θέλετε να χάσουμε το χρόνο μας, να θυσιάσουμε το χρόνο μας, αλλά με αυτόν τον τρόπο, αλλά πραγματικά είναι κρίμα για τους υπόλοιπου βουλευτές από άλλε χώρε. Κύριε Τέρη Κάμπρα, θα συνεχίσετε με αυτό το πολιτικό διάλογο. Ναι, αλλά θεώρησα ότι μπορούσα να πω κάτι για το χρονοδιάγραμμα. Και αυτό θέλω να κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα που συζητάμε εδώ είναι πολύ σοβαρό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα πρόγραμμα και πρέπει να έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό και αντιτίθαμε σε αυτά που έλεγε η συνάδελφος. Αν το θέμα είναι σημαντικό και είναι, προκειμένου να αποφύγουμε πολιτικούς ελιγμούς, πρέπει ακριβώς να αδιαφορήσουμε για το πότε υπάρχουν εκλογές. Να έχουμε το δικό μας το ρυθμό. Ό,τι και αν συμβεί εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όποιες είναι οι άλλες ημερομηνίε και τα ραντεβού που υπάρχουν. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ που μας βοηθάτε. Πραγματικά. Συνεπώς, η κυρία Αλβιών. Μπορείτε κι εσείς να είσαστε εξίσου πολύτιμοι και να μας βοηθήσετε. Ναι. Διαφωνώ με την πρόταση της κυρίας Σεστάρας. Καθημερινά υφίστανται έξωση οικογένειες στην Ισπανία επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν την, υπόθηκα δάνειά τους. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ήταν θύματα της απάτης με τις προνομιακές μετοχές. Όλα αυτά από το 2011 δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε περισσότερο. Ούτε μπορεί να δίνουμε την εντύπωση ότι μας απασχολούν πιο πολλοί εκλογές στην Ισπανία από ότι οι πολίτες που θίστανται τις εξώσεις ή για εκείνους οι οποίοι είναι θύματα απατών. Δεν είναι αυτή η εικόνα που θέλουμε, ότι μπορούμε να αφήσουμε εξωτερικά στοιχεία να καθορίσουν το έργο μας. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δουλέψουμε, για να προχωρήσουμε με τα ψηφίσματα που θέλουμε να προχωρήσουμε και θεωρούμε σωστά. Οπότε το χρονοδιάγραμμα που θα υιοθετήσουμε είναι εκείνο το οποίο θα μας επιτρέψει με τη συζήτηση που θα γίνει να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πριν τα Χριστούγεννα δηλαδή. Πρόεδρος, Σολεδάδ, θες και εσύ να παρέμβεις. Για το χρονοδιάγραμμα μόνο. Είναι σαφές νομίζω. 24 Ιουλίου, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όπως νομίζετε ότι θα λειτουργήσει καλύτερα το πράγμα. Τίποτα άλλο δεν είχα να πω. Μόνο αυτό. Ρώσα. Θέλω να επαναλάβω ότι δεν είναι τυχαίο που η πρόταση αυτή ψηφίσματος ε, μας τη φέρατε τώρα και με αυτόν τον τρόπο κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γι' αυτό και η Ισπανική κυβέρνηση, αν θέλετε να μπούμε στην ουσία, έχει εφαρμόσει διάφορα συγκυριακά και διαφορετικά μέτρα για να μην γίνει άλλο αυτό που έγινε με κώδικα καλής για τις κατοικίες, για την, ε, το ότι δεν γίνονται πληρωμές, με νομοθεσία, με ρυθμίσεις και επίσης όσον αφορά τις προνομιακές. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι τυχαίο που ήρθε τώρα το θέμα αυτό. Όχι για να ανταποκριθούμε στο αίτημα των καταγγέλλοντος, που συμφωνώ. Όντως πρέπει να απαντήσουμε στον καταγγέλλοντα. Αλλά πιστεύω ότι έρχεται τώρα αυτό το θέμα εδώ εξαιτία άλλων πολιτικών συμφερόντων. Δεν είναι τυχαίο, Σεσίλια. Τι να κάνουμε που γίνεται τώρα ενώ έχουμε εκλογέ ε, την Νοεμβρία. Δεν τον Δεν είμαστε ε, αθώοι, κανένα από εμά. Υποστηρίζω του, τα θύματα από τι εξώσει από τις προνομιακέ κτλ. Αλλά να μην υπάρχουν και άλλα συμφέροντα, όπως και εσεί δώσατε την απόψή σα, δίνω εγώ και τη δικιά μου, ότι υπάρχουν εδώ πέρα πολιτικά κριτήρια και βάσει αυτών έγινε εδώ πέρα αυτό το θέμα σήμερα. Αν ήταν ε, τόσο σημαντικό, τότε δεν θα συζητάγαμε έναν 24 που το καλοκαίρι θα το αφήναμε για το Σεπτέμβριο. Εγώ ειλικρινά, αν σκεφτόμαστε τα θύματα από τις υποθήκες και τα προνομιακέ τις προνομιακές μετοχές, τότε να μην τα συνδέουμε όλα αυτά με τις εκλογές. Δεκέμβριο, εντάξει, Δεκέμβριο, κανένα πρόβλημα. Για να υποστηρίξουμε τα ε, συμφέροντα των πολιτών. Και μην σκεφτόμαστε το χρονοδιάγραμμα της Ισπανίας. Βλέπετε μόνο Ισπανοί μιλάμε εδώ, οπότε δεν είναι τυχαίο. Πρόεδρος, ωραία. Δεν έχω άλλους ομιλητές. Έχω δύο προτάσεις τώρα. Ή που τηρούμε το αρχικό χρονοδιάγραμμα που σας είπα, προθεσμία δηλαδή για τροπολογίες 24 Ιουλίου και έγκριση στην Επιτροπή μας το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο πιθανώ στην Ολομέλεια, αυτή είναι η μία εναλλακτική. Η άλλη εναλλακτική είναι προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, η 10η Σεπτεμβρίου, μετά δηλαδή τις διακοπές, ψηφίζουμε στην Επιτροπή μας τον Οκτώβριο και το Δεκέμβριο κατά πάσα πιθανότητα στην Ολομέλεια. Ποιο από τα δύο προτιμάτε. Προτιμάτε την πρώτη εναλλακτική λύση ή τη δεύτερη. Ποιο είναι υπέρ της πρώτης εναλλακτική λύσης. Δηλαδή προθεσμη 24 Ιουλίου για τροπολογίες. Και ποιο είναι υπέρ της εναλλακτική 2. ΕΛΚ, Άλτε, η FTD, το μισό η FTD. Κοιτάξτε, πρέπει να μετρήσω τα χέρια, έτσι. Ακούστε. Ωραία, με τις κάρτες σας. Βάλτε στο μηχάνημα τις κάρτες σας ηλεκτρονικά. Θα δούμε. Λοιπόν, εναλλακτική λύση 1. Ποιοι είναι υπέρ της πρώτης εναλλακτικής λύσης ή κατά της πρώτης λύσης. 24 Ιουλίου. Ναι ή όχι. Ψηφίζετε ανάλογα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη σοφορίας. Έντεκα ψήφοι υπέρ. Δώδεκα κατά. Έντεκα υπέρ, δέκα κατά. Άρα τον Ιούλιο. Παρακαλώ κύριε Μάτο. Κοιτάξτε. Όποιος πρότεινε να αναβληθεί η ψηφοφορία για το Σεπτέμβριο, τώρα ψήφισε υπέρ του να γίνει τον Ιούλιο. Δεν είναι καταπληκτική η επιτροπή μας. Πρόεδρος, κοιτάξτε, καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα της Επιτροπής Αναφορών. Επαναλαμβάνω. Καλώ ήρθατε στην πραγματικότητα. Οι καταστάσει αλλάζουν ε, ταχύτατα. Ο Ενρίκο. Μία διόρθωση. Είπατε ότι η Άλντε έκανε κάτι. Όχι. Ο Ενρίκε Καλβέτ που δεν δέχεται εντολές. Εγώ καταψήφισα. Γιατί για να κάνω σωστά τη δουλειά μου ήθελα περισσότερο χρόνο. Δεν το έκανε αυτό η Άλντε, ο Ενρίκε Καλβέτ. Οπότε περνάμε στο επόμενο θέμα της μέρης διάταξης, που είναι η παρουσίαση. Κοιτάξτε τώρα, μπορείτε όλοι να χαλαρώσετε και να ακούσετε το τμήμα πολιτικής ΣΥ, το οποίο θα μας παρουσιάσει το θέμα της υιοθεσίας ε, χωρίς συνένεση. η Κλέα Φέντον Γκλίν που είναι λέκτορας ε, επινομικών θεμάτων στο κολέγιο Kings του Λονδίνου. Καλησπέρα, λέγομαι Κλέα Φέντον Γκλίν. Είμαι λέκτορας ε, στο νομικό τμήμα στο King's College. Έχω πρώτο πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Αδελαίδας στην Ισπανία και ένα μάστερ σε νομικά θέματα από την Οξφόρδη και ένα διδακτορικό για τα δικαιώματα των παιδιών από το Cambridge. Όλη μου η εργασία και μετά το διδακτορικό είναι το θέμα της υιοθεσία και οι διαφορετικοί τρόποι με τον οποίο τα κράτη-μέλη ασχολούνται με την προστασία των παιδιών. Η Επιτροπή μου ζήτησε να ασχοληθώ με το θέμα που θέτουν μια σειρά αναφορές σε σχέση με τον αυξανόμενο αριθμό παιδιών που τα αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες προστασίας των παιδιών στην Αγγλία και κατόπιν δίδονται για υιοθεσία. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει συνένεση για αυτήν την υιοθεσία γονική. Προς το συμφέρον των παιδιών δεν απαιτείται αυτή η συνένεση. Έχετε ένα αντίγραφο της έκθεσής μου που μπαίνει σε πολλές λεπτομέρειες αλλά θα κάνω μια σύντομη επισκόπηση του συστήματος ε, υιοθεσία στην Αγγλία και την Ουαλία. Πρώτον, το σύστημα της υιοθεσία δεν μπορεί να διαχωριστεί από το σύστημα προστασίας των παιδιών με βάση των αγγλικών νόμων. Τρεις αρχές. Πρώτα απ' όλα είναι αρχή του καλού για το παιδί. Πάντα το πρωταρχικό, το μόνο είναι το συμφέρον του παιδιού. Δεύτερη είναι η αρχή του να μην γίνονται καθυστερήσει. Διότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά το μέλλον ενό παιδιού μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ε, στην καλή ποιότητα ζωή του. Και τρίτον, η αρχή τη μη παρέμβαση. Ότι πρέπει να παρεμβαίνει το κράτο ή μια οικογένεια μόνο αν είναι αναγκαίο με βάση το άρθρο 8 τη ε, Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βάσει θεμελιωδών δικαιωμάτων, συγγνώμη. Για να ξεκινήσει η διαδικασία υιοθεσία πρέπει να υπάρχουν δύο κριτήρια. Πρώτο είναι το κατόφλι ζημίας. Δηλαδή το δικαστήριο πρέπει να θεωρεί ότι το παιδί μπορεί να βλαβεί ή υπάρχει κίνδυνος να βλαβεί. Και είναι πολύ ευρία η έννοια της βλάβης, της ζημίας. Για παράδειγμα μπορεί να είναι κακομεταχείριση, προβλήματα στην υγεία, την ανάπτυξη, μπορεί να υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση, συναισθηματική κακοποίηση και επίσης ε, προβλήματα μπορεί να έχει στην ε, φυσιολογική, την κοινωνική, εκπαιδευτική κλπ. ανάπτυξή του. Αυτή είναι η ευρεία απόπειρα ορισμού του τι σημαίνει ζημία. Αλλά για να ε, αντισταθμιστεί αυτό πρέπει να είναι σοβαρή ζημία, ουσιώδη ζημία. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι προβλήματα που δημιουργούνται λόγω ανεπάρκειας ε, των ανθρώπων και της ασταθούς συμπεριφοράς του. Ένα από τα βασικά θέματα που αναφέρουν διάφορες αναφορές είναι τι κίνδυνος υπάρχει στο μέλλον να υποστεί ζημία το παιδί. Αυτό μπήκε στην ομοθεσία για τα παιδιά το 1999 επιτρέπει στις τοπικές αρχές να αναλάβουν πρωτοβουλία να δράσουν, δηλαδή να πάρουν ένα παιδί και να αναλάβουν την επιμέλειά του, αν υπάρχει βάση για να πιστέψει κανείς ότι στο μέλλον θα υποστεί ζημία. Βέβαια το θέμα κλειδί είναι πώς γίνεται αυτή η αποτίμηση, σε ποια βάση επιτρέπεται το δικαστήριο να θεωρήσει ότι υπάρχει κίνδυνος. Ότι πληρούνται δηλαδή αναγκαίες ε, προϋποθέσεις και υπάρχουν δύο τεστ που κάνουν οι αρχές. Πρώτον, βέβαια πρέπει να δούμε το ποιο είναι πιο πιθανό για το αν υπάρχουν οι συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε μια τέτοια πράξη. Υπάρχουν συνθήκες τέτοιες, μπορεί να αποδειχθεί ότι ισχύουν και κατόπιν εξετάζουμε το ενδεχόμενο μελλοντική ζημίας. Πρώτα λοιπόν το δικαστήριο πρέπει να εξετάσει τους ισχυρισμούς για το πώς έχει τρέχουσα κατάσταση ή τι έχει συμβεί στο παρελθόν που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι θα υποστεί στο μέλλον ζημία το παιδί. Και μετά θα πρέπει να δουν τι μπορεί να σημαίνει η ζημία αυτή στο μέλλον. Και εδώ βέβαια είναι χαμηλότερη πιθανότητα που πρέπει να ισχύει. Η λέξη για παράδειγμα ενδεχόμενο είναι πιθανό σημαίνει ότι υπάρχει ουσιώδης πιθανότητα για, σε σχέση με τη φύση και τη σοβαρότητα της μελλοντική ζημίας. Αν αυτό το κατόφλιο ζημίας θεωρηθεί ότι έχει ξεπεραστεί, τότε τίθεται το θέμα της γονικής ε, συγκατάθεσης. Είτε ο γονέας πρέπει να εγκρίνει την υιοθεσία ή μπορεί να παραβλεφθεί η έλλειψη έγκρισης. Το δικαστήριο δεν μπορεί να παραβλέψει εάν δεν θεωρήσει ότι ισχύουν οι συνθήκες για να παραβλέψει την ανάγκη γονικής συγκατάθεσης. Οποιαδήποτε απόφαση για την υιοθεσία λαμβάνει υπόψη, όπως είπαμε, το καλύτερο συμφέρον, ε, το καλό του παιδιού. Όταν καταλήξει το δικαστήριο ότι είναι προς το καλύτερο συμφέρον του παιδιού να δοθεί προς υιοθεσία, αυτό σημαίνει ότι το καλό του παιδιού σημαίνει ότι πρέπει να παραβλεφθεί η ανάγκη για γονική συγκατάθεση. Όταν καθορίζουμε εάν το καλό του παιδιού προϋποθέτει υιοθεσία πρέπει να ληφθούν υπόψη μια σειρά από παράγοντες που τους βλέπετε εδώ για παράδειγμα το καλό του παιδιού για όλη του τη ζωή συμπεριλαμβανομένης και της επίδρασης που θα έχει ότι θα αφαιρεθεί από την οικογένειά του και τη διακοπή οποιονδήποτε σχέσεων ε, ενδεχομένως με την αρχική του οικογένεια. Ο όρος ότι ε, πρέπει να υπάρχει αυτή η ανάγκη να παραβλεφθεί με βάση την ομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σημαίνει ότι τα δικαιώματα, του παιδιού, τα δικαιώματα των γονέων συγγνώμη, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη με, τρόπο που να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας. Αν βλέπουμε τώρα τι γίνεται για, την, ε, για να παραβλεφθεί η γονική συνένεση. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες αγνόησης ας πούμε ή, ε, για να θεωρηθεί ότι δεν είναι αναγκαία η γονική συνοχή. Βέβαια υπάρχει επικάλυψη και ορισμένα κράτη χρησιμοποιούν δύο ή τρία από αυτά τα κριτήρια. Η πρώτη ομάδα είναι αν δεν αναγκαία η συγκατάθεση γιατί έχει εγκαταλειφθεί το παιδί ή δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ορισμένα κράτη θέτουν χρονικά όρια που πρέπει να περιμένουν δηλαδή οι αρχές πριν θεωρηθεί ότι ισχύει αυτό το κριτήριο. Δεύτερο κριτήριο, δεν είναι αναγκαίες η κατάθεση γιατί είδε είναι κακή η συμπεριφορά των γονέων ή έχουν αφαιρεθεί τα γονικά του δικαιώματα ή υπάρχει συγκεκριμένη συμπεριφορά των παιδιών για παράδειγμα ε, κακομεταχείριση ή αμέλεια που θέτουν κινδύνο την υγεία των παιδιών. Ο τρίτος λόγος είναι αν οι γονείς έχουν ε, αρνηθεί συγκατάθεση ε, χωρίς να έχουν αιτιολογήσει τους λόγους αυτούς ή αν πρέπει να παραβλεφθεί για να εξυπηρετηθούν τα καλύτερα συμφέροντα του παιδιού. Αυτό είναι με βάση και τις αρχές των ΗΕ ότι τα συμφέροντα του παιδιού. Είναι το άρθρο 21 αυτό τη σύμβαση για τα παιδιά των ΗΕ που λέει ότι το συμφέρον του παιδιού είναι το πρωταρχικό. Τώρα υπάρχουν μηχανισμοί χωρίς συνένεση σε όλες τις χώρες μέλη. Αλλά ο νόμος στην Αγγλία οδηγεί στις περισσότερες υιοθεσίε. Την 21η Μαρτίου 2014 βλέπουμε ότι 5.050 παιδιά είχαν υιοθετηθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό είναι αύξηση σε σχέση με το 2013 κατά 26% και 58% σε σχέση με το 2010. Και 96% αυτών των υιοθεσιών έγιναν χωρίς γονική συνένεση. Ωστόσο, ωστόσο. Ναι, μεν υπάρχει συνεχής αύξηση. Είναι σημαντικό να δούμε ότι τους τελευταίους 6 μήνες έχει υπάρξει άξιο σημείο τη μείευση των υιοθεσιών. Και αυτό βασίζεται σε μία απόφαση του εφετείου διότι το δικαστήριο ήταν ιδιαίτερα επικριτικό έναντι του τρόπου λειτουργίας των τοπικών αρχών στην Αγγλία και είχε σοβαρές ανησυχίες και δισταγμούς για τον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν το θέμα της υιοθεσία χωρίς συγκατάθεση. Και είπαν ότι τα δικαστήρια πρέπει να είναι πιο προσεκτικά και να μελετήσουν πολύ πιο αυστηρά όλες τις αποφάσεις των τοπικών αρχών για να καθίσταται σαφές γιατί είναι αναγκαία η υιοθεσία προς το καλύτερο συμφέρον των παιδιών αντί να επιλεγούν άλλε εναλλακτικέ λύσεις. Πολλά έχουν υποθεί για τους στόχους που θέτει για υιοθεσίε για τις δημόσιες αρχές στην Αγγλία. Λίγο πριν ε, την έγκριση του νέου νόμου υπήρχε στόχο στο Ηνωμένο Βασίλειο να αυξηθούν οι υιοθεσιε κατά 40 50% και μέχρι το 2005 είχε υπάρξει αύξηση 38% έκτοτε, συγκεκριμένα με το 2006 δεν υπάρχουν επίσημοι στόχοι, αλλά έχουμε δει ότι ο Πρωθυπουργό και ο Υπουργό που είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά είπαν ότι δεν θα αρκεστούν σε αύξηση απλώς θέλουν να υπάρξει ε, βελτίωση των παιδιών, του αριθμού των παιδιών που υιοθετούνται από την επιμέλεια των δημοσίων αρχών. Αλλά πρέπει να τονίσω ότι η επίπτωση του καθορισμού στόχων δεν σημαίνει ότι παίρνουμε περισσότερα παιδιά, παίρνουν οι αγγλικές αρχές περισσότερα παιδιά από τα σπίτια τους. Αλλά αυτό που έχουν ως στόχο αυτή η στόχη είναι ότι εάν θεωρηθεί ότι τα παιδιά πρέπει να αφαιρεθούν από το γονικό περιβάλλον, πρέπει να υιοθετούνται ταχύτατα προ το συμφέρον των παιδιών, όπω είπαμε και προηγουμένω, για να γίνει σεβαστή και η αρχή τη μη καθυστέρηση. Στο τέλο τη έκθεσή μου, κάνω μια σειρά από συστάσει και προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και προ το Ηνωμένο Βασίλειο. Μία από τις κυριότερες προς την Ένωση είναι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ιδιαίτερα κατευθυντήριες γραμμές για περιπτώσεις διαμεθοριακών υιοθεσιών, δηλαδή να δίνεται κατάλληλη πληροφόρηση που πρέπει να είναι διαθέσιμη προς τις κυβερνήσεις και προς αυτούς που ασχολούνται με τον ε, τομέα αυτό για να καταλαβαίνουν καλύτερα τα διαφορετικά συστήματα που υπάρχουν. Επίσης, πολλές φορές δεν ενημερώνονται οι κυβερνήσεις ότι κάποιος υπηκός του σε άλλη χώρα έχει ε, γίνει αντικείμενο επιμέλειας από τις αρχές άλλου κράτους. Επίσης συστήνουμε να υπάρξει και να ενθαρρυνθεί περισσότερη κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων και να γίνει περισσότερη έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή. Για το Ηνωμένο Βασίλειο οι οικογένειες πρέπει να συνεχίσουν να δέχονται βοήθεια, ούτως ώστε η υιοθεσία να είναι μόνο τελευταία καταφυγή. Αν ένα παιδί δεν μπορεί με κανένα τρόπο να παραμείνει στο σπίτι του με την οικογένειά του και πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Περισσότερα πρέπει να κάνουμε και για να βελτιώσουμε και την κατάσταση των παιδιών που είναι υπό δημόσια επιμέλεια και να δούμε ποιες άλλες εναλλακτικέ λύσεις πρέπει να βρεθούν πέρα από την υιοθεσία για τα παιδιά που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Γιατί βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση των παιδιών που είναι υπό δημόσια επιμέλεια. Δεν είναι καθόλου καλή αυτή η κατάσταση. Και είπαμε ότι ναι μεν δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το πολιτιστικό και γλωσσικό ε, υπόβαθρο του παιδιού, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη γενικά ε, το, ε, το από πού προέρχεται. Εγώ σας ευχαριστώ για αυτές, αυτές τις τόσο αναλυτικές πληροφορίες που μας δώσατε είναι πραγματικά αυτό που μας δίνεται μια εξαιρετική μελέτη, όχι μόνο για την Επιτροπή Αναφορών, αλλά και για ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, γιατί τώρα αρχίσαμε σιγά σιγά και βήμα προς βήμα να αντιμετωπίζουμε αυτό το πολύ ευαίσθητο και σοβαρό θέμα της προστασίας των παιδιών και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρ ε, Φέντον Γκλίν, ε, για αυτήν την εξαιρετική παρουσίαση του θέματος. Στρέφουμε τώρα στην Πατρίσια Ντελούκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα της δώσω το λόγο έτσι ώστε ε, να έχουμε και τη δική της θέση σχετικά με αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω ευχαριστεί τη δόκτωρα Κλέρε Φέντον Γκλίνε για αυτήν την μελέτη η οποία σίγουρα Indeed, adoption without η οποία βεβαίως ε, ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμη και οπωσδήποτε θα βγει ιδιαίτερως ε, και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερόμαστε στα δικαιώματα του παιδιού και φυσικά εμείς έχουμε προσυπογράψει και την Χαρτά Εθνών για την εναλλακτική επιμέλεια και προστασία των παιδιών. Εμείς έχουμε φυσικά και νομοθεσία για τις υιοθεσίε, αλλά πρόκειται για αρμοδιότητα που δεν είναι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, ε, αλλά ε, η οποία υπόκειται σε κάποιες ε, συνθήκες όπως ε, η διεθνή ε, Συνθήκη για τις ε, Υιοθεσίες και η σχετική σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οπωσδήποτε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις εξουσίες που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Η Κομισιόν μπορεί να παρέμβει μονάχα εάν ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, ε, παραβιάζεται. Έχουμε βεβαίως έναν κανονισμό που αφορά την απομάκρυνση παιδιού από έναν γονιό. Έχουμε κάποιες περιπτώσεις αμφισβητούμενης επιμέλειας, αλλά ε, σε, περίπτωση, ε, ε, σε τέτοιες περιπτώσεις μάλλον έχουμε δύο ή περισσότερα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι και η δική σας Επιτροπή Αναφορών έχει μελετήσει περιπτώσεις παιδιών με διπλές υπηκότητες, αλλά το γεγονός ότι εμπλέκονται παιδιά με διπλές ας πούμε ε, υπηκότητες ή που έχουν μια υπηκότητα και έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα από αυτήν που είναι τη συνήθους τους διαμονής. Παρόλα αυτά ε, η περίπτωση δεν γίνεται υποχρεωτικά ε, διασυνοριακή. Είναι ακόμα εθνική περίπτωση. Να σας πω επίσης ε, ότι δεν υπάρχει από άποψη ευρωπαϊκής νομοθεσίας κανονισμός ο οποίος αναφορά το δικαίωμα επίσκεψης, τη συχνότητα των επισκέψεων κτλ. Όλα αυτά ε, ε, σε περιπτώσεις μοιρασμένης επιμέλειας καθορίζονται από τις ε, οι επιμέρους νομοθεσίες των κρατών μελών. Έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Ενδεχομένως γνωρίζετε ότι εμείς βρισκόμαστε σε φάση τροποποίησης αναμόρφωσης του κανονισμού Βρυξέλλες 2 ε, και ε, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω τροπολογιών ε, και επομένως όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ακούμε σήμερα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα και για μας. Πρόεδρος, Μα εδώ έχουμε ένα εξαιρετικά καλό παράδειγμα διαθεσμικής, διοργανικής ε, συνεδρίας, ε, συνεργασίας. Νομίζω ότι μπορεί να είναι μια εξαιρετικά επικοδομητική διαδικασία και οπωσδήποτε ε, δίνει τροφή για σκέψη, για διάλογο, για περαιτέρω συνεργασία και βεβαίως αυτό εν ώψη της διερευνητικής αποστολής ε, που θα κάνουμε αργότερα ε, στη διάρκεια του τρέχοντος έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, πραγματικά πολύ σωστή χρονική στιγμή που γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, η κυρία Ντανόκα θα ξεκινήσει το γύρο των αγορητών. Μόλις χτες έλαβα μια επιστολή από ένα ζευγάρι εθωνών που ζουν στην Σκοτία. Έχουν ένα παιδάκι τριών μηνών που ε, είχε ψηλό πυρετό, το πήγαν το μωράκι στο νοσοκομείο και οι γιατροί Ε, υπέθεσαν ότι το παιδί έπεσε και αυτό προκάλεσε το ψηλοπυρετό. Οι γονείς είπαν ότι όχι δεν συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά αυτό αποτέλεσε αιτία να τους αφαιρέσουν το παιδί. Δεν το δέχτηκαν οι γονείς βέβαια ε, και προφανώς ε, οι γιατροί θεώρησαν ότι υπήρχε παραμέληση ανηλίκου. Ε, και μάλιστα κάπου το ανέφερε και η κυρία Φέντον Γκλίν ε, ε, εκεί που λέτε για κακή μεταχείριση, για παραμέληση ανηλίκου λοιπά. Όμως οι γονείς ήταν πραγματικά σοκαρισμένοι, δεν, ενδεχομένως τα προβλήματά τους προέκυψαν για, από ελληπή γνώση της αγγλικής γλώσσας αλλά οι γιατροί επέμειναν ότι το παιδί αρρώστησε ε, γιατί έπεσε και αποφάσισε ε, οι γιατροί να καλέσουν τις ε, ε, υπηρεσίες ε, τις κοινωνικές ε, και να απομακρύνουν το παιδί από την οικογένεια αυτό το ζευγάρι των Εστονών. Παρόμοιες επιστολές λαμβάνω και από άλλους Λετονούς, Λιθουανούς, Εστονούς που ζουν και έχουν παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν επανειλημμένα αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Καταλαβαίνω και αυτό που είπε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, κατανοώ τις ε, συστάσεις ε, της δόκτωρος Φέντον Γκλίν, γιατί οι συστάσεις σας δεν είναι και ανατρεπτικές και επαναστατικές. Είστε επιστήμον και όχι πολιτικός, αλλά πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι το πρώτο και μεγαλύτερο προβλήματα είναι ε, αυτό ακριβώς το θέμα της υιοθεσία χωρίς συγκατάθεση που είναι μια διαδικασία που πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε και συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Επιτροπή Αναφορών. Αυτοί πρέπει ίσως να αναλάβουν ε, οι, οι ντόπιοι ε, βουλευτές λοιπά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την λέκτορα Φανενγκλίν. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη της. Όλοι θυμόμαστε πόσο φορτισμένες ήταν οι ακροάσεις της Επιτροπής Αναφορών που ακούσαμε διάφορες οικογένειες, διάφορους γονείς και η μελέτη αυτή ακριβώς δείχνει πού βρισκόμαστε νομικά και πρακτικά. Είναι πολύ χρήσιμο. Και θα είναι πολύ χρήσιμο να ενημερώσουμε και την ερευνητική αποστολή. Τώρα για τόσο ακούσαμε εμείς, οι πολιτικοί έχουμε την ευθύνη να μην προσπαθούμε να είμαστε ριζοσπαστικοί όταν πρόκειται για την προστασία του παιδιού. Ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι προστατεύονται παρκώς τα παιδιά και ότι το σύστημα και οι έλεγχοι του συστήματος γίνονται καλά σε όλες τις χώρες, όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Ένα από τα στοιχεία κλειδί που θέσατε πάντως είναι η ιδέα αυτή της υιοθεσίας χωρίς συγκατάθεση είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε σε όλα τα νομικά συστήματα των χωρών μελών. Εφαρμόζεται περισσότερο ή λιγότερο συχνά στις διάφορες χώρες μέλη, υπάρχει όμως σαν νομική δυνατότητα. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε ο έλεγχος του συστήματος πώς γίνεται. Και σε αυτό θα βοηθήσει και η ερευνητική αποστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως ε, βουλευτής από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτή την ερευνητική αποστολή, πολύ σωστά. Θα ακούσουμε τις εμπειρίες των βουλευτών που θα πάνε και θα δούνε πώς έχει η κατάσταση στην πραγματικότητα. Όλοι οι φορείς πάντως και στην Αγγλία και στην Ουαλία και στις τοπικές αρχές θα συνεργαστούν. Θα ήταν ενδιαφέρον να κοιτάξουμε λίγο κατά πόσο υπάρχουν ε, περισσότερες πιέσεις τα τελευταία χρόνια προς τις υπηρεσίες προστασίας των παιδιών εξαιτία των οικονομικών περικοπών. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και εκείνες προστασίας των παιδιών, εγώ πιστεύω ότι πιέζονται εξαιτία των περικοπών στον προπολογισμό. Ενώ δεν θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι καλό να δούμε τι ισχύει. Καλή είναι και η ενημέρωση όσον αφορά το τι ισχύει νομικά, ποιες είναι οι τελευταίες αποφάσεις που έχουν γίνει, για να δούμε πώς ενημερώνεται η Βρετανική νομοθεσία. Και σίγουρα να δούμε αν ελέγχεται καλά το σύστημα. Τέλος, τι κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το στοιχείο κλειδί είναι στην αναθεώρηση της, του κανονισμού Φρυξέλλες 2. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όχι μόνο αυτή η μελέτη, αλλά και τα αποτελέσματα της διερευνητικής αποστολής, να δούμε πώς βλέπουν τα διασυνοριακά ζητήματα. Στην αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2 υπάρχει αυτό το στοιχείο. Είναι σαφές ότι ο κανονισμός αυτός είναι το νομικό πλαίσιο, το καταλληλότερο μέσα στο οποίο τίθενται όλες οι αποφάσεις. Πάντως θα είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Έτσι ώστε όλοι να μπορούν να δουν ποιος κάνει τι και πώς. Τέλος. Αυτά τα ζητήματα είναι συναισθηματικά φορτισμένα και δύσκολες περιπτώσεις. Κάθε φορά που φεύγει ένα παιδί από τους γονείς του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό γίνεται για τους σωστούς λόγους, για το καλό του παιδιού δηλαδή. Δεν λέω ότι είναι τέλειο το σύστημα. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε πάντα ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα στο σύστημα. Πάντως θα ήθελα να αποφύγω, πώς να το πω, κάνω έκκληση. Όπως ελπίζουμε, και το λέω ως Βρετανίδα, Ελπίζω ότι οι υπόνοιες αυτές που υπάρχουν για τις Βρετανικές τοπικές αρχές δεν ισχύουν, δεν ευσταθούν. Ότι δηλαδή έχουμε στόχο κάποιες συγκεκριμένες εθνικότητες. Δεν το πιστεύω. Και ελπίζω όταν η ερευνητική αποστολή πάει στον Ηνωμένο Βασίλειο, ελπίζω να μην πάει με προκαταλήψεις κατά των Βρετανών. Πρέπει να δούμε πραγματικά τι γίνεται και πώς λειτουργεί το σύστημα και τι μαθήματα μπορεί να πάρει κανείς. Γιατί ναι, ίσως να έχουμε μεγαλύτερα νούμερα και η μελέτη σας εξηγεί το γιατί, αλλά υπάρχουν θέματα και σε άλλες χώρες μέλη. Και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να πάρουμε τα μαθήματά μας και αυτά είναι ισχύουν όχι για μία χώρα, αλλά για την κατάσταση συνολικά. Συστήνω λοιπόν ότι δουλειά έχει γίνει μέχρι τώρα από τους συναδέρφους να ληφθεί υπόψη. Και σε προσωπικό επίπεδο σας λέω ότι είμαι σε καλύτερη κατάσταση σήμερα από ότι όταν τέλειωσε η ακρόαση που είχαμε με τις οικογένειες, γιατί πραγματικά νιώθα τότε εξαντλημένη, έπρεπε να πάω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο να συνέλθω πρέπει και εκείνοι να νιώθουν ότι τους έχουμε ακούσει, ότι έχουμε λάβει υπόψη μας το όσα έχουν πει και ότι εμείς τους εκπροσωπούμε δίκαια. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Αυτό που λέτε είναι ακριβώς αυτό που όλοι νιώσαμε μετά από αυτήν την τόσο λεπτή και βέστητη συνεδρίαση. Η κυρία Μαγκίνες τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή που ήταν τόσο σαφής και σε βάθος και ευχαριστώ και για τις συστάσεις γιατί λέει κάποια πράγματα που το αισθηκτό μας λένε μερικές φορές αλλά τώρα το βλέπουμε και σαν συμπέρασμα της μελέτης αυτής. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα βέβαια. Εγώ, ως τη μεσολαβητής από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Προστασία των Παιδιών, Όντω και εγώ πήρα πάρα πολύ στα σοβαρά όλε αυτέ τι. σε όλα αυτά που μα είπαν οι γονεί στην ακρόαση, οι οποίοι ένιωσαν ότι δεν τηρούνται τα δικαιώματά του δεν προστατεύονται όταν πρόκειται για υιοθεσίε. Το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί αυτό το μηχανισμό πιο συχνά από ότι άλλε χώρε μέλη. Αυτό είναι σαφές. Θα ήθελα να ξέρω τώρα για τι δικαστικέ αποφάσει. Όταν μα απαντήσετε, μπορείτε να μα αιτιολογήσετε καλύτερα τις δικαστικές αυτές αποφάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί τα νούμερα και να μας πείτε το κοινωνικό σύστημα που προσανατολίζεται. Ξέρετε ότι πολλοί από μας πήγαμε σε συνάντηση στο Ηνωμένο Βασίλειο που οργανώθηκε από τη Σλοβακική Πρεσβεία. Ήταν πολύ σημαντική και η έκθεσή σας νομίζω το λέει. Όσοι ήμασταν εκεί και πήραμε το λόγο, είδαμε ότι το νομικό σύστημα είναι διατεθειμένο να ακούσει τις απόψεις και τις εμπειρίες άλλων ε, χωρών. Θα ήθελα λοιπόν να δω το άρθρο 15 να χρησιμοποιείται καλύτερα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και το 56 του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Είχα την αίσθηση ότι κάποιες πρεσβείες στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα βοηθούν καλύτερα τους δικούς τους πολίτες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γονείς που έχουν ε, στερηθεί τα παιδιά τους γιατί το βρετανικό σύστημα τα έχει δώσει για αναδοχή γεωθεσία. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει και το πρόβλημα το γλωσσικό που είναι ένα επιπλέον εμπόδιο για τους γονείς αυτούς. Πάντως, αυτό που πρέπει να λέμε και να ξαναλέμε είναι ότι πάντα το συμφέρον του παιδιού προέχει είναι κάτι που δεν ορίζεται βέβαια πάντα με σαφήνεια και η ερμηνεία είναι μερικές φορές υποκειμενική. Πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε όμως και νομικά τι σημαίνουν οι όροι και οι λέξεις. Ποιες είναι οι επιλογές που έχουν τα παιδιά και οι οικογένειες που βρίσκονται σε δυσκολία. Να στηρίξουμε την οικογένεια, τη στηρίζουμε αρκετά σε όλες τις χώρες και το τελευταίο σχόλιο είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτό πρέπει να το δούμε για όλες τις χώρες μέλη και να μην επικεντρωνόμαστε σε μία μόνο. Πρέπει επίσης να δούμε οι οικογένειες που τελικά στερούνται το παιδί τους, τι είναι προτιμότερο, ε, προστασία του παιδιού σε κάποια παράδειγμα ανάδοχη οικογένεια ή υιοθεσία. Και στη χώρα μου την Ιρλανδία είχαμε προβλήματα με την υιοθεσία και τώρα έχουμε φτάσει στις συνέπειες. Κάποιοι ενήλικες για παράδειγμα τώρα διαπιστώνουν ότι οθετήθηκαν με το ζόρι στο παρελθόν. Πολύ ευαίσθητο θέμα, πολύ λεπτό. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα και η Επιτροπή Αναφορών, η οποία πολύ σωστά κάθισε και άκουσε τις λιβερές αυτές τις ιστορίες. Όταν έχει πάει η οθεσία στον Ηνωμένο Βασίλειο ένα παιδί, εμείς πώς θα επιστρέψουμε το παιδί στην οικογένειά του. Είναι πολύ θλιβερό, αλλά είναι η πραγματικότητα παππούδε. Έχω μια τέτοια περίπτωση για δύο αγόρια όταν κάποιο μάθει την ιστορία είναι πραγματικά πολύ θλιβερό να βλέπει τι γίνεται. όμω δεν μπορώ να παρέμβω νομικά. Αυτό πάντως που πρέπει να κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε σε διάφορα επίπεδα και το κάνουμε στην Επιτροπή Αναφορών. Χρειαζόμαστε όμως και άλλους συναδέρφους ώστε να ακουστεί πιο πολύ και στην Ολομέλεια αυτό το ζήτημα και σε όλες τις χώρες μέλη. Να προβληθεί, να μιλήσουμε πιο πολύ για τα θέματα προστασίας του παιδιού τι γίνεται στις χώρες μέλη μας, τι συμβαίνει, τα συστήματα προστασίας του παιδιού τι κάνουν. Υπάρχει κάποια κοινή δομή παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λόγο επίσημη επ' αυτού, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή δομή μεταξύ όλων των χωρών και να αναγνωρίσουμε ότι κάποιες χώρες μέλη, και τις αναφέραμε εδώ, κατηγορούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά ένα παιδί που γεννιέται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι Βρετανός πολίτης, οπότε αναγκαστικά υποβάλλεται στο σύστημα προστασία των παιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου και θα συμφωνήσει και συνάδελφο ότι το σύστημα θέλει να βελτιωθεί. Δεν θέλουμε να βρεθεί ένα παιδί σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση επειδή δεν ε, παραβήκαμε έγκαιρα. Εδώ χρειάζεται η σοφία του Σολομόντος για να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει. Ε, δεν την έχουμε όλοι. Πρέπει να εμπιστευτούμε το σύστημα προστασίας του παιδιού, ότι λειτουργεί καλά, αλλά βέβαια αν έχουμε αφιβολίες πρέπει να το ψάχνουμε. Και χαίρομαι που ακούω ότι υπάρχει μια ομάδα εργασίας για τα θέματα προστασίας του παιδιού και πολύ θα ήθελα να μπορέσω να έχω επαφές με αυτήν την ομάδα εργασίας για να βοηθήσουμε κι εμείς. Η έκθεσή σας αποτελεί μια πολύ καλή βάση για όλους μας προκειμένου να προχωρήσουμε. Σας είπα πριν και το άρθρο 15 όταν ακούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με την αναθεώρηση που θα γίνει στο Brussels 2 και το άρθρο 56 επίσης και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε για να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια. Οι πρεσβείες μας επίσης έχουν να παίξουν ρόλο. Πρόεδρε, ο δικό σα ρόλο τώρα στην Επιτροπή Αναφορών, εσεί πρέπει να εξετάσετε όλε τι αναφορέ και σα εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σα. Ξέρω ότι οι άνθρωποι ήρθαν εδώ, άνοιξαν την καρδιά του σε εμά και εμεί ίσω δεν μπορέσουμε να του δώσουμε την απάντηση που χρειάζονται. Αλλά πρέπει να του πούμε ότι μα έκαναν να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και ελπίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τι μελλοντικέ ίσω οικογένειε, όχι αυτέ που έχουν ήδη υποφέρει, αλλά τις μελλοντικέ βάσει των συστάσεων που έχουμε και βάσει των όσων έχουν να προσθέσουν οι συνάδελφοι. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας το συμφέρον του παιδιού πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πολύ σε βάθος ανάλυση της κατάστασης και σας ευχαριστώ επίσης που τονίσατε ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε εσφαλμένες προσδοκίες. Δεν είμαστε δικαστήριο, δεν είμαστε δικαστές, είμαστε εκπρόσωποι των πολιτών της Ένωσης. Προσπαθούν να βρούμε μη δικαστικές ε, λύσεις για αυτές τις τρομερά δύσκολες και λεπτές καταστάσεις. Και μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε πολλές δραστηριότητες ε, που προγραμματίζουμε το φθινόπωρο μαζί με την Νομική Επιτροπή για παράδειγμα κοινή ακρόαση πριν την αναθεώρηση του κανονισμού Φρυξέλλες 2 έχουμε ομάδες εργασίας, έχουμε διερευνητικές επισκέψεις και φυσικά με χαρά θα συνεργαστούμε μαζί σας κυρία Μαγκίνες για το θέμα αυτό η ομάδα εργασίας ούτε ξέρουν ποιος θα συμμετάσχει αλλά θα είναι ένα μέλος από κάθε ομάδα και θα ορίσουν τον πρόεδρό τους και φυσικά μπορείτε πάντα, είστε ευπρόσδεκτοι, μπορείτε πάντα να ε, λάβετε μέρος. Ο κύριος Μαριάς. Α συγχαρώ τη δόκτωρα Κλέρ Φέντον Γκλίν για την ε, πολύ καλή δουλειά που έκανε και για την παρουσίασή της και να πω ότι οι υιοθεσίες χωρίς συνένεση είναι ένα θέμα οικογενειακού δικαίου και θεωρητικά αν το σκεφτεί κανείς θα μπορούσε να πει ότι δεν αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αφορά την ε, λειτουργία της, επομένως ενδεχόμενα δεν αφορά και την Επιτροπή Αναφορών. Το γεγονός βεβαίως ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο κανονισμό ε, Βρυξέλλες 2 που μάλιστα θα αναθεωρηθεί δείχνει ότι υπάρχει ένα στοιχείο ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και κυρίως αυτό αφορά την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων Δηλαδή είναι ένα διαδικαστικό θέμα για το πώς θα εκτελούνται, θα αναγνωρίζονται οι δικαστικές αποφάσεις μεταξύ των κρατών μελών. Όμως από τις ακροάσεις που είχαμε, αλλά και από τη μελέτη, προκύπτει ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα και στην ε, Μεγάλη Βρετανία ε, και στην Γερμανία για υιοθεσίες χωρίς συνένεση και είδαμε περιπτώσεις που είχαν έρθει εδώ και μας κατήγγυλαν και για το Γιούγκενταμ και για την ε, Αγγλία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα των δύο κρατών. Αν αφορούσε μόνο τους Γερμανούς πολίτες, προφανώς. Αλλά είδαμε ότι υπάρχουν μερικά στοιχεία που για μένα δεν είναι τυχαία. Ότι αρκετοί από τους αναφέροντες και παραπονούμενους τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων ή και οι δύο δεν είναι πολίτες των συγκεκριμένων κρατών. Δηλαδή δεν είναι πολίτες της Αγγλίας ή πολίτες της Γερμανίας, αλλά είναι πολίτες άλλων κρατών μελών. Και μπαίνει ένα ερώτημα αν η μεταχείριση που έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες στην Αγγλία ή στη Γερμανία απέναντι στους πολίτες που δεν είναι Άγγλοι ή Γερμανοί είναι ίδια με αυτή απέναντι σε πολίτες άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μήπως υπάρχει μια συνεχής εφαρμογή διαφορετικών κριτηρίων και συμπεριφοράς. Άρα μήπως έχουμε μια διοικητική πρακτική των συγκεκριμένων υπηρεσιών πρόνοιας στην Αγγλία και στη Γερμανία που είναι διακριτική, discriminatory απέναντι στους πολίτες άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εδώ αμέσως Υπάρχει ένα ζήτημα εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου, είναι η παραβίαση και η διακριτική μεταχείριση της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, διότι οι πολίτες άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα είναι και πολίτες της Ένωσης. Και αν υπάρχει διακριτική μεταχείριση είναι σίγουρα θέμα εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου, επομένως είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν να δει αν γίνεται παραβίαση συστηματική του ευρωπαϊκού δικαίου και επομένως να προσφύγει κατά των συγκεκριμένων κρατών. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Και ανέφερε η συνάδελφος ότι υπήρχαν δύο συμπολίτε της που συνέβη να πάνε το παιδί του στο νοσοκομείο και επειδή το ερώτημα είναι επειδή ήταν λετονοί τους φέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο ή θα, θα έκαναν το ίδιο και αν είχαν απέναντί τους δύο γονείς που ήταν Άγγλοι ή Σκοτσέζοι. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να δούμε. Και επειδή βλέπουμε πολλές τέτοιες καταγγελίες, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα από πρώτης απόψεως, αλλά θα το διερευνήσουμε βεβαίως και στις επισκέψεις που θα κάνουμε στην Αγγλία και ίσως και στις άλλες περιπτώσεις, να δούμε αν υπάρχει τέτοια διακριτική μεταχείριση. Και θα πείτε, μα γιατί να υπάρχει τέτοια διακριτική μεταχείριση. Ποιο είναι το κίνητρο. Γιατί να υπάρχει μια τέτοια εφαρμογή. Εγώ βλέπω στην έκθεση, εδώ που μας ε, ε, έχετε μοιράσει, ε, στη σελίδα 22, βλέπω ότι υπάρχει και κάποιος λόγος ενδεχόμενα. Λέει εδώ στην έκθεσή της η κυρία Φέντον Γκλίν ότι, και θα το διαβάσω στα αγγλικά, ότι η κυβέρνηση ε, ότι υπάρχει ένα report that called on που καλούσε τις τοπικές αρχές και την κυβέρνηση να αυξήσουν ριζικά τον αριθμό υιοθεσιών στην Αγγλία. Είναι μια κατεύθυνση να αυξηθούν οι υιοθεσίες. Και στην επόμενη σελίδα, στη σελίδα 23, διερευνά αν υπάρχουν και κίνητρα, bonuses τα οποία δίνουν οι τοπικές, οι local authorities για να έχουμε αύξηση των υιοθεσιών. Επομένως είναι μια στρατηγική ενός κράτους και παίρνουν και μπόνους οι ίδιοι οι υπάλληλοι των τοπικών, των local authorities για να αυξήσουν τις υιοθεσίες και τυχαίνει να είναι υιοθεσίε που γίνονται σε πολίτες που δεν είναι πολίτες της Αγγλίας αλλά άλλων κρατών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ ανοίγει μια ολόκληρη υπόθεση που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά το Ευρωκοινοβούλιο, αφορά την Κομισιόν, η οποία και στην άλλη συζήτηση που είχαμε για τον Γιούγκενταμ μα έλεγε ότι δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον όρο ότι οι εμπλεκόμενοι είναι πολίτε άλλων κρατών και του αφαιρούνται τα αστικά δικαιώματα επιμέλεια των παιδιών. Αλλά και η μεταχείριση των ίδιων των παιδιών τα οποία και αυτά είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια ότι έχουν την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να είναι κάτω από 18 ετών, αλλά προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, είναι λοιπόν αρμοδιότητα αυτή. Και βλέπουμε στην επόμενη σελίδα, σελίδα 25 και 26 υποθέσεις όπου συγκεκριμένα κράτη διαμαρτύρονται. Λάτβια, ε, Βουλγαρία, Σλοβακία, Τσεχία κλπ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμείς έχουμε αρμοδιότητα ως Επιτροπή Αναφορών να παρεμβαίνουμε όχι για να λύσουμε ένα οικογενειακό ζήτημα, γιατί αυτό είναι δύσκολο, αλλά για να αντιμετωπίσουμε μια διοικητική πρακτική που μπορεί να είναι και discriminatory, διακριτική, εις βάρος πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως αυτό το θέμα είναι τεράστιο και χαίρομαι που ήδη αποφασίσαμε να ιδρύσουμε αυτό το working group στο πλαίσιο της Επιτροπής μας. Θα κάνουμε και την επίσκεψη στην Αγγλία και νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι πλέον επιτάπητος και πρέπει να τα δούμε από μια άλλη διάσταση. Για να καταλάβουμε κι εμείς για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η συμπεριφορά από τις αρχές στην Αγγλία και στη Γερμανία που είναι αρμόδιες για τις υιοθεσίε. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά. Ποιο είναι, ποια είναι η βαθιά σκέψη. Τι κρύβεται πίσω. Και Πώς τυχαίνει πολλές καταγγελίες να είναι από πολίτες που δεν είναι πολίτες είτε στην Αγγλία είτε στη Γερμανία. Αυτά λοιπόν τα θέματα νομίζω είναι σημαντικά. Εγώ να σας συγχαρώ ξανά για την ε, πολύ καλή δουλειά που κάνατε. Ε, είχα μια πρώτη ευκαιρία να ρίξω μια ματιά, αλλά προφανώς διαβάζοντας περισσότερο θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε. Επομένω, νομίζω ότι η συζήτησή μας έχει πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία Μαγκίνης, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή μπορεί με την παρουσία της και το ρόλο της να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην όλη υπόθεση για να μπορούμε και εμείς ως Επιτροπή Αναφορών να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό ζήτημα που είναι πλέον φλέγον ζήτημα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Soledad, Ευχαριστώ πολύ, Soledad. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Πολλά ακούσαμε ήδη από τους συναδέρφους και θέλω να πω ότι η εργασία αυτή είναι μια πολύ καλή βάση για αυτό το θέμα. Με ευθύ με υπεύθυνο τρόπο μπόρεσε να συμπεριλάβει αυτά τα οποία και εμείς ε, λέμε κατά τη διάρκεια όλης αυτής της ε, θητείας. Και αναφέρει και πολλά από αυτά που και εμείς στην ομάδα εργασίας έχουμε πει. Πρόκειται για διάφορες χώρες, με διαφορετικό τρόπο διαπιστώνουμε το φαινόμενο αυτό και κατά πάσα πιθανότητα έχει να κάνει και με την ερμηνεία του τι είναι η προστασία του ανήλικα. Πρέπει να δούμε όμως αν υπάρχουν διακρίσεις τελικά και αν έχει να κάνει με την προέλευση ή όχι του ατόμου ή πρόκειται για τη διαφορετική απλώς ερμηνεία όπως σας είπα και πριν που η κάθε χώρα βλέπει διαφορετικά αυτό το θέμα. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες, σε διάφορα μέτρα. Τα πρέπει όλα να τα μελετήσουμε, να τα αναλύσουμε για να καταλήξουμε σε ποια κοινωνική πολιτική στήριξη της οικογένειας και του παιδιού είναι καλύτερη στις διάφορες χώρες. Γιατί πολλές φορές καταλήγουμε σε αναγκαστικές συμπεριφορές και όχι σε πραγματική κοινωνική πολιτική προς το συμβαίνον της οικογένειας και του παιδιού. Αυτό πρέπει να το δουν οι πυρογνώμονε, βέβαια στην ε, ψυχολογία, στην ομάδα εργασία, Λαμβάνουν υπόψη μα και αυτό προκειμένου να μας εξηγήσουν τι είναι καλύτερο να κάνουμε. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό σαν μας είπατε, ως βάση για το έργο μας. Θα ανταλάβουμε υπόψη μας. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού που έχει επικυρωθεί σχεδόν από όλα τα μέλη και αν μη τι άλλο να προβάλλουμε τα προβλήματα αυτά των παιδιών που δεν έχουν φωνή εδώ, που δεν είναι εδώ. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ο Πέτρο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την κυρία Φέντσον Γκλίν για την παρουσίαση. Στην Επιτροπή Αναφορών τα θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι πάντα πολύ περίπλοκα. Και χρειαζόμαστε και την άποψη των νομικών και η μελέτη σας διευκρινίζει το θέμα, παρουσιάζει όλες τις περιπτώσεις, θα μας βοηθήσει στη δουλειά μας. Δεύτερον, Βέβαια, πολύ συχνά, όπως είπε και κάποιος προηγούμενος, συζητούμε τα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συζητήσουμε και μια προφορική ερώτηση. Αλλά έχω κάποια ερωτήματα για να καταλάβω καλύτερα. Πάντα όταν ακούω ότι έγινε μία υιοθεσία χωρίς τη γονική συγκατάθεση αισθάνομαι άσχημα γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιστραφεί. Όπως είπατε και στην ε, μελέτη σας, ε, μπορεί τα αίτια να είναι η κακομεταχείριση, η παραμέληση. Ξέρετε όμως ότι μπορεί να έχουν προβλήματα και οι γονείς. Ε, μπορεί σε αυτή τη φάση να πηγαίνουν άσχημα τα οικονομικά τους ή να περνάνε κάποια κρίση και σε δύο-τρία χρόνια να βελτιωθεί η κατάσταση των γονιών. Αν όμως το παιδί του το έχουν πάρει και έχει υιοθετηθεί χωρίς την άδειά του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορούν να ε, επιδιώκουν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Δεν θα ήταν καλύτερα να αναλάβουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες ε, το παιδί και να μην υπάρξει υιοθεσία χωρίς την ε, έγκριση των γονέων. Γιατί αλλιώς πάντα αισθάνομαι άβολα όταν βλέπω τέτοια πράγματα. Άλλο ερώτημα. Γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τη διευρυμένη οικογένεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις το παιδί που είχε, ε, είχε αν, ανέτρεφε, ανέτρεφε μόνη η μητέρα, πατέρθηκε κάποιον άλλον, το έδωσε η υιοθεσία. Γιατί δεν σκεφτήκαμε τον βιολογικό πατέρα και δεν μπόρεσε να παίξει το ρόλο του. Και η διευρυμένη οικογένεια. Ξέρετε ότι πολλές φορές ε, είναι σε θέση οι παππούδες και οι γιαγιάδες ε, να παίξουν το ρόλο τους. Γιατί τι γίνεται με τα δικαιώματα, με το καλό του ίδιου του παιδιού. Όπως είπατε, οι 60-70% των ε, υιοθεσιών γίνονται μεταξύ ενός και τεσσάρων ετών. Αλλά τα παιδιά μεγαλώνουν. Δεν τους ρωτάμε, δεν τα ρωτάμε τη γνώμη τους. Αποφασίζουν άλλοι για αυτά, ακόμη και αν είναι μεγαλύτερα, για την τύχη τους. Και αυτό με ανησυχεί. Γιατί θεωρώ, λοιπόν, ότι από κοινού πρέπει στην Ευρώπη να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε αυτή η χωρίς συγκατάθεση η υιοθεσία πρέπει να είναι απόλυτη εξαίρεση για να μην υπάρξει καμία παρανόηση. Σε αυτήν την επίσκεψή μας στην Αγγλία θα συμμετάσχουν και Άγγλοι βουλευτές, αλλά όχι ως ε, επίσημοι συμμετέχοντες. Μπορούν να παρευρεθούν και μάλιστα μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει και οι βουλευτές ε, της χώρας όπου πηγαίνουν να συμμετέχουν. Αυτά ήταν τα ερωτήματά μου, γιατί πραγματικά με ανησυχεί το, το θέμα αυτό εντάξει υπάρχουν, υπάρχουν ε, και διαφορετικές ερμηνείες για το τι σημαίνει παραμέληση. Ε, ξέρετε ότι αυτά τα οποία γίνονται ορισμένε φορέ στη μία άκρη τη Ευρώπη μπορεί να θεωρηθούν παραμέληση στην άλλη άκρη τη Ευρώπη. Τέλο. Κάτι με το οποίο συμφωνώ απόλυτα από αυτά που είπατε. 200%. Χρειαζόμαστε περισσότερη επικοινωνία με τα κράτη-μέλη. όταν οι γονείς είναι από διαφορετικά κράτη-μέλη πρέπει να βοηθούν και τα κράτη-μέλη. Γιατί πολλά προκύπτουν από παρεξηγήσεις. Δεν καταλαβαίνει ο ένας ε, τη νομική κατάσταση του άλλου. Ο καθένας θεωρεί ότι αυτό που ισχύει στο κράτος του ισχύει και στα άλλα κράτη-μέλη. Φυσικά δεν ισχύει. Αλλά είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, προχωρεί η ενοποίησή μας. Πρέπει λοιπόν από κοινού να επιχειρήσουμε, να λύσουμε ε, τις διαφορές μας και να επιτύχουμε συμβιβασμού. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Η κυρία Πιτέρα, τελευταία ομιλήτρια για το θέμα αυτό και θα, θα μιλήσουμε μετά για την έκθεση από τη Στρογγυλή Τράπεζα για το Δικαίωμα των παιδιών. Παρακαλώ. Α, και η κυρία Ντανόκα. Ωραία, και εσείς, βέβαια, βεβαίω, τελευταία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε μάλλον για αυτήν την ε, μελέτη και την παρουσίαση που μας κάνατε. Ε, είμαι ευγνώμων κυρίως όσον αφορά την, τα συμπεράσματά σας ε, σχετικά με την διασυνοριακή ανταλλαγή συμπερασμάτων και την αύξηση της γνώσης των διαδικασιών και της ευαισθητοποίησης λοιπόν που πρέπει να προκύψει. Ε, τα δικαιώματα των γονιών είναι συγκεκριμένα και δεν είναι δυνατόν ε, να απομακρύνουν τα παιδιά ε, χωρίς λόγο. Υπάρχουν πολλές καταχρήσεις και καταχρηστικές συμπεριφορές από τους από τις κοινωνικές υπηρεσίες ε, ε, και πολλές φορές ε, δεν είναι σωστές οι πληροφορίες που έχουν. Από την άλλη πλευρά οι γονείς προσπαθούν πάντα να βρουν κάποιες δικαιολογίες, πολλές φορές ψεύτικες. Επίσης, οι πήκοοι άλλων χωρών ε, οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες ε, θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να κάνουν μια προσπάθεια προσαρμογής. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει και οι κοινωνικές υπηρεσίες να γνωρίζουν και κάποιες παραδόσεις ενδεχομένως των χωρών από τις οποίες προέρχονται. Η Ισράσου Μαγκίνες αναφέρθηκε στην ανάγκη ε, συνεργασίας και διπλωματικής ε, ε, και συνεργασίας μέσω διπλωματικών αντιπροσώπων και τα λοιπά. Επίσης, τα κέντρα υποστήριξης των ε, ε, οικογενειών ας πούμε ε, θα πρέπει να συνεργάζεται, να συνεργάζονται. Στην περίπτωση της Πολωνίας η συνεργασία του συγκεκριμένου φορέα με την πολωνική πρεσβεία είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλη μείωση των αριθμών των υιοθεσιών και των, της απομάκρυνσης παιδιών από Πολωνούς υπηκόους. Περισσότερη βοήθεια, καμιά φορά και ηλική βοήθεια, ε, που θα ε, πρέπει να δίνεται από το κέντρο γίνεται πιο αποτελεσματική σε συνεργασία με την ε, πρεσβεία. Υπάρχουν και κάποιοι φραγμοί οι οποίοι καμιά φορά θολώνουν την κρίση και επομένως εμποδίζουν την πλήρη αντικειμενικότητα. Πάντως, σίγουρα η ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και η ανταλλαγή πληροφοριών ε, είναι κάτι πάρα... Είναι απαραίτητο. Η κυρία Ντανόκα. Θα κάνω κι εγώ μια επιπλέον παρατήρηση που προκύπτει από τη συζήτηση. Διαβάζουμε εδώ αυτήν την ε, ε, έκθεση, την μελέτη της κυρίας Φέντον Γκλίν, την οποία ευχαριστούμε, αλλά διαρκώς αναφέρεστε ε, στον κανονισμό Βρυξέλλες 2, προστασία της οικογένειας κτλ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχουμε και την βασική αρχή, το βασικό δικαίωμα ε, της ελεύθερης κυκλοφορίας ε, των εργαζομένων και των πολιτών. Φανταστείτε λοιπόν Λετωνούς, Εστονούς ή οπουδήποτε αλλού, αλλά κυρίως πολίτες της Ανατολικής ε, Ευρώπης και σας ευχαριστώ που κάνετε συγκεκριμένη αναφορά στη σελίδα 25 ε, αναφέρεστε σε ε, ε, καλά στοιχειοθετημένες περιπτώσεις οι οποίες έχουν μελετηθεί ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να σας πω λοιπόν έλεγα ε, ότι ε, οι πίκοοι αυτών των ανατολικών χωρών πολλές φορές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν έρχονται ας πούμε στη χώρα αυτή οι γονείς και να δουλέψουν και μετά έχουν πρόβλημα με τα παιδιά τους στη χώρα αυτή, στην ουσία παραβιάζεται και το δικαίωμα που έχουν σε αναζήτηση εργασίας αλλού. Πρόεδρος, ακούσατε λοιπόν αγαπητή δόκτωρα Γκλίν ε, τις απόψεις και τις ερωτήσεις ε, των μελών της Επιτροπής ε, και θα σας δώσω δύο λεπτά έτσι ώστε να απαντήσετε. Πολλές είναι οι ερωτήσεις οι οποίες τέθησαν, δεν θα μπορέσω να τις απαντήσω μέσα σε δύο λεπτά, θα προσπαθήσω. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι να υπογραμμίσουμε τον λόγο για τον οποίο όλες οι χώρες έχουν ένα σύστημα υιοθεσία ε, χωρίς συγκατάθεση ε, και αυτό γίνεται οπωσδήποτε ε, προς το συμφέρον του παιδιού για περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει το παιδί να απομακρυνθεί από το παιδί σε περίπτωση ας πούμε συναισθηματικής παραμέλησης ή φυσικής σεξουαλικής ε, βίας. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ε, αναφέρθηκε ότι και από την πλευρά τους οι κοινωνικές υπηρεσίες μερικές φορές καταχρώνται των δυνατοτήτων που τους δίνει ο νόμος και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, μονάχα όταν ε, το παιδί βρίσκεται ε, υπό αστυνομική επιμέλεια διαφοροποιείται η κατάσταση διαφορετικά και θα πρέπει εντός 72 ώρων η υπόθεση να φτάσει ενώπιον του δικαστηρίου σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία. Βεβαίως οι γονείς λέτε μπορεί και να αλλάξουν. Βεβαίως μπορεί να ε, ανακτήσουν ε, μια διαφορετική, ε, καλύτερη κατάσταση. Και βεβαίως το σημαντικό είναι για μας όμως, για, για, τους, για τις κοινωνικές υπηρεσίες, το παιδί όσο γίνεται πιο γρήγορα να πάει σε ένα ασφαλές περιβάλλον και γνωρίζουμε ότι σε περιπτώσεις ε, παιδιών που έχουν ζήσει πολλά χρόνια σε ιδρύματα ξέρουμε ότι είναι επιρρεπή ε, σε με, μετέπειτα εγκλισμό σε φυλακή και τα λοιπά. Από, του, από τον ε, πληθυσμό των σοφρονιστικών ιδρυμάτων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει περάσει από τέτοιου είδους ιδρύματα. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε φυσικά. τώρα, τα studies of social ε, Τα μέτρα λιτότητας ε, αν και η μετακίνηση των ε, εργαζομένων γονιών λόγω των μέτρων λιτότητας. Ναι, βεβαίως αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά καταλαβαίνετε ότι λόγω και των μέτρων λιτότητας πολλές φορές οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες δεν έχουν τα κονδύλια τα οποία είναι απαραίτητα ή ακόμα και τους ε, ανθρώπινους πόρους έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν σωστά όλες τις ε, περιπτώσεις. Ε, θέλετε να πείτε κάτι άλλο σχετικά με το... Ε, είχα κάνει μια συγκεκριμένη ερώτηση για τις δικαστικές διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι και διμερώς μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, λέει η Πρόεδρος, ε, διμερώς νομίζω είναι καλύτερο να το λύσετε το θέμα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να σας ευχαριστήσω, ε, δόκτωρα Φέντον Γκλίν, για την μελέτη σας. Αυτή η έρευνα που κάνατε είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και ε, ενδεχομένως και η γραμματεία θα σας απευθύνει αργότερα ε, και κάποια ερωτήματα εάν και, κατα... εάν και εφόσον προκύψουν. Τώρα ε, έχουμε και την έκθεση της κυρίας Μαγκίνες μετά από την εκδήλωση της Σλοβενικής Πρεσβείας στο Λονδίνο 17 Μαΐου έγινε αυτή η ε, συνάντηση και νομίζω ότι πολλοί θα είναι οι αυτοί που ενδιαφέρονται να πάρουν το λόγο, αλλά παρακαλώ να μην μακρηγορήσετε. Κυρία Μαγκίνες, διαμεσολαβήτρια, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ήταν θαυμάσια αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστώ την Σλοβακική Πρεσβεία και όλους και το Διεθνές Νομικό Κέντρο για την Προστασία των Παιδιών και των Νέων. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση. Υπογράμμισε πολλά από τα θέματα που θίξαμε και μόλις τώρα. Ότι δηλαδή οι Βρετανικές αρχές αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά για πολίτες άλλων κρατών διαφορετικά. Η εντύπωση, λέω, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα, δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Αλλά όλοι οι νομομαθείς λοιπόν εκεί, πρώτα απ' όλα να πω ότι ο Ζε Μάθιου Θόρπ, ο οποίος είναι σύμβουλος Σλοβακικής Πρεσβείας, ήταν συντονιστής Σερ James Μάμπι, που είναι αρμόδιος στο ανώτατο δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας για θέματα οικογενειακού δικαίου έκανε μια πολύ καλή παρουσίαση της κατάστασης συμπεριλαμβανομένων και πολλών λεπτομεριών όπως αυτές που αναφέρατε ιδίω για το θέμα αυτό ποιο είναι το καλό του παιδιού σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επίσης είπε ότι έχουν ευθύνη και οι δικαστές και οι κοινωνικές υπηρεσίες να ενημερώνουν ε, τις προξενικές υπηρεσίες όταν ε, τίθενται θέματα άλλων πολιτών άλλων κρατών για να λάβουν την αναγκαία βοήθεια. Και το αποδέχεται το δικαστικό σύστημα στην Αγγλία και την Ουαλία ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα γι' αυτό. Επίσης ε, η εφαρμογή του άρθρου 15 του Βρυξέλλες 2 για την μεταφορά υποθέσεων σε άλλα κράτη-μέλη και γι' αυτό πρέπει να γίνουν παραπάνω πράγματα και καλωσορίζω την πρόθεση της Κομισιόν να ασχοληθεί. Επίσης είχαμε μια, μια παρουσίαση από την ε, δικαστή ε, κυρία Μπλακ για μεμονωμένες περιπτώσεις που μπορούν να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη αλλά πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της ε, αλλαγής δικαιοδοσίας Άρα πρέπει να απλοποιηθεί το άρθρο 15, να το δούμε αυτό. Ορισμένοι από τους παρόντες συζητήσαμε με τους αναφέροντες αλλά και η υπηρεσία μου επειδή είμαι διαμεσολαβήτρια συζήτησε με τους αναφέροντες οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να πω ότι έχουν κάθε καλή διάθεση να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα αυτό να συνεργαστούν περισσότερο Είπαμε ότι θα συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Να υπάρξει λοιπόν αυτή η αύξηση συνεργασίας για να βοηθήσουμε τους πολίτες που εγκαθίστανται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι χωριστά τα δικαστικά συστήματα, γιατί κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του, αλλά πολλά μπορούμε να κάνουμε για να υπάρξει περισσότερη δικτύωση, για να υπάρξει περισσότερη αλληλοκατανόηση. Και υπάρχει καλή θέληση και βούληση να επιτευχθεί αυτό. Ίσως μπορούμε να παίξουμε εμείς ως Επιτροπή Αναφορών καταλητικό ρόλο, να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή σχόλια στη διάθεσή σας, ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς το λόγο από αυτού. Η κυρία Πιτέρα, παρακαλώ. Ήμουν παρούσα σε αυτή τη συνάντηση το Μάιο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πολύ επικοδομητική. Να προσθέσω ότι η κατάσταση αλλάζει ριζικά και ταχύτατα απτά στο σύστημα προστασίας παιδιών. Τον Ιανουάριο 2004 υπήρξε αυτή η απόφαση ορόσημων. στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα ε, οι κοινωνικές υπηρεσίε που ασχολούνται με τα θέματα αυτά είναι πολύ πιο προετοιμασμένες και τα προξενία των ε, χωρών των οποίων οι πολίτες εμπλέκονται ενημερώνονται για επικείμενες διαδικασίες ενημερώνονται για το ενδεχόμενο παρουσίας των κοινωνικών λειτουργών στα δικαστήρια. Οπότε, έχει αλλάξει η κατάσταση. Παλιά, κατά την ακροαματική διαδικασία, οι γονείς των παιδιών δεν μπορούσαν να μιλήσουν στον τύπο όσο εκκρεμούσαν οι υποθέσεις. Τώρα έχει αλλάξει η κατάσταση. Ξέρω την κατάσταση γιατί στη χώρα μου, στην Πολωνία, έχουμε περιπτώσεις όπου επέστρεφαν από την Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο επίκοοι μας και μίλαγαν στον τύπο γιατί δεν μπορούσαν να μιλήσουν όσο ήταν στις χώρες αυτές. Αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον. Αυτή λοιπόν η συνάντηση στο Λονδίνο που διοργάνωσε η Σλοβακική Πρεσβεία ήταν πολύ επικοδομητική, και αποδεικνύεται ότι αν υπάρχει βούληση πάντα υπάρχει τρόπος. Και νομίζω ότι είχαμε και πολύ καλή συνεργασία με διάφορα προξενικά γραφεία διαφόρων κρατών μελών της Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να αποδώσουν, μπορούν να βοηθήσουν αν δεν υπάρχει αρνητική ε, συναισθηματική φόρτιση, αν υπάρχει καλή διάθεση για να επιληθούν τα πραγματικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτρα Γιά. Ευχαριστώ. Και εγώ είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή την εκδήλωση. Να σας δώσω μια πολιτική εκτίμηση από πλευράς μου. Είναι πολύ ευνοϊκή η κατάσταση. Πρέπει να δράσουμε για το θέμα αυτό. Αναμφίβολο είναι αυτό. Τα θέματα έχουν τεθεί και διαπιστώσαμε για θέματα περιπτώσεων υποθέσεων στην Αγγλία διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να μιλήσουν μαζί μας. Γιατί στο παρελθόν τα κράτη-μέλη έλεγαν όχι, έχω το δικό μου σύστημα και ο καθένας, το κάθε κράτος μέλος, έλεγε το δικό μου είναι το καλύτερο, αφήστε με ήσυχο. Αυτό ίσχυε και για τη Γερμανία και τη Δανία. Στην Αγγλία για πρώτη φορά είδαμε να έχει αλλάξει το κλίμα, να λένε χρειαζόμαστε διάλογο, γιατί δεν είναι όλα στο συμβαίνουν ε, τα καλύτερα. Αυτό το κλίμα θα έλεγα είναι λοιπόν ένα παράθυρο ευκαιρίας για να προχωρήσουμε το θέμα αυτό, να το συζητήσουμε, γιατί τα κράτη-μέλη θέλουν να βοηθήσουν. Είναι μοναδικό θα έλεγα, ή σχεδόν μοναδικό, είχε αλλάξει πολύ η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτήν την εκδήλωση. Είχα τις αμφιβολίες μου αν θα είχε έννοια, αλλά έμαθα πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και συμμετείχατε στο Λονδίνο. Μπράβο, πολύ καλό. Να διατηρήσετε τα διάφορα συμπεράσματα, να τα κρατήσετε, θα είναι σίγουρα πολύ χρήσιμα για όλους μας όταν θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα κάποια στιγμή. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Το επόμενο θέμα είναι η γνωμοδότηση για την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια συνολική αντιμετώπιση της μετανάστευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ψήφισμα της 17ης Δεκεμβρίου που μας πέρασε, το ΕΛΚ ζήτησε από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να αξιολογήσει τις σημερινές πολιτικές όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο και να πάει στην Ολομέλεια μέχρι τα τέλη της χρονιάς αυτής μέσω μιας έκθεσης πρωτοβουλίας. Στόχος της έκθεσης αυτής λοιπόν είναι με συνολικό τρόπο να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις πολιτικές και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του ασύλου και της μετανάστευσης να ασχοληθεί με θέματα όπως είναι η διεθνής προστασία, η έλεγχη στα σύνορα, η κοινή ευθύνη, η χρηματοδότηση και προκειμένου να καταλήξει και σε συστάσεις. Έχουμε δύο συντάκτες, η κυρία Έγγελ από του Σοσιαλιστές και η κυρία Μετσόλα από το ΕΛΚ. Και εγώ είμαι σκιώδης εισηγείται, από πλευράς του Άλντε, των φιλελεύθερων. Άρα με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Και για μας είναι η κυρία Αλέν Μίτσι, η συντάκτρια γνωμοδότηση. Σα δίνω και το λόγο κυρία Μίτσι, λοιπόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, δυστυχώς και πολύ επίκαιρο. Είναι κάτι που μας απασχολεί όλους για να συντάξω τη γνωμοδότησή μου περιοριστικά βέβαια από το μέγεθος της γνωμοδότησης και συνεπώς δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω όλες τις πληροφορίες, όλες τις ιδέες και όλα τα σημαντικά θέματα που θα ήθελα να συμπεριλάβω όπως για παράδειγμα το πόσο πολλά είναι τα παιδιά το οποίο διασχίζουν την ε, Μεσόγειο, πόσο μεγάλη σημασία έχει να υπάρξει κάποια τροποποίηση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, η δράση της Frontex, ο Τρίτον, ούτε μπόρεσα να τα βάλω όπως πρέπει, αλλά έτσι από το παράθυρο θα προσπαθήσω να συμπληρώσω αυτά τα μέτρα στη συνέχεια. Είμαστε Επιτροπή Αναφορών, οπότε ο κύριος στόχος μου ήταν να ασχοληθώ με τον μεγάλο αριθμό που μας υποβάλλουν οι πολίτες. Έπρεπε να το λάβω αυτό υπόψη μου. Και επικεντρώθηκα λοιπόν σε τέσσερα κυρίως σημεία οι αναφέροντες εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για τον μεγάλο αριθμό θανάτων μεταξύ των ανθρώπων που προσπαθούν να διασύσουν τη Μεσόγειο. Και ακριβώς επειδή οι τραγωδίες αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες και πολύ συχνά ε, βλέπουμε να περνάνε τη Μεσόγειο, γι' αυτό λέμε σαν συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει παρατηρητής, αλλά πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να εγκρίνει το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, μετανάστευση. Αναφέρομαι επίσης τις ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των ε, ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δράσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται και να ενισχύονται. Επίσης η πολιτική ασύλου πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια σε διεθνείς προδιαγραφές στον οποίο έχει καταρτιστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω επίσης ότι οι χώρες μέλη πρέπει να εγκρίνουν ε, παρόμοιες πολιτικές και πρακτικές που να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια. Και λέμε επίσης ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την εφαρμογή των αρχών που έχουν να κάνουν με τη μεταναστευτική μας πολιτική. Τρίτον, Αναφέρομαι στην αποτελεσματικότητα, αλλά και ε, στις αδικίες που υπάρχουν μέσω του συστήματος του Δουβλίνου. Άρα πρέπει να βρεθούν νέες λύσεις, γιατί αυτές που έχουμε μέχρι τώρα δεν είναι αποτελεσματικές. Το σύστημα του Δουβλίνου βάζει υπερβολικά μεγάλο βάρος πάνω σε ορισμένες χώρες μέλη, κυρίως αυτές που βρίσκονται στην περιφέρεια. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως. Τέταρτον, αναφέρομαι στην έλλειψη πραγματικής πολιτικής μεταναστευτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε λοιπόν να ενισχυθεί η μεταναστευτική πολιτική και να ενισχυθεί το θεματολόγιο που αναφέρεται στην μετανάστευση. Μιλάμε τώρα για αλληλεγγύη και καταμερισμό ευθυνών. Όμως, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια τα οποία καθυστερούν τη διαδικασία. Άρα η Ευρώπη χρειάζεται μια συνολική πολιτική μετανάστευσης και ασύλου που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και αξίες και αρχές πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επίσης να σχεδιάσουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι και νομίζω ότι κάποιες χώρες μέλη πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για το μέλλον της μετανάστευσης. Μέχρι τώρα συλλέγονται στοιχεία, δεδομένα από διάφορες υπηρεσίες, μη οργανώσεις, εθνικές αρχές κλπ. Όμως δεν υπάρχει ένας κοινό τρόπος για να κυκλοφορούν τα στοιχεία αυτά. Γι' αυτό και ζητούμε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συλλογής δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εκπονεί εκθέσεις τακτικά, που θα ενισχύσει το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση κρίσεων. Θα διαχειρίζεται κρίσεις. Πρέπει να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε όλα τα δεδομένα για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Τέλος, ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό προσπαθώ να είμαι σύντομη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά δεν θα προχωρήσουν γρήγορα. Πρέπει οι λύσεις μας να είναι μακροπρόθεσμες και να αντιμετωπίσουμε και τις ρίζες της μετανάστευσης. Να διασφαλίσουμε ότι η πρόοδος και η καλή εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής θα λειτουργήσουν. Αλλά να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η αναχώς αυτή η έξοδος από τις χώρες προέλευσης τόσο πολλών ανθρώπων. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ χωρών μελών. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να πολεμάει και ελπίζω ότι θα βρούμε καλές λύσεις διάρκειας. Προσβλέπω σε επικοδομητικό διάλογο μεταξύ μας. Σίγουρα θα καταφέρουμε να έχουμε μια πολύ καλή έκθεση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η τώρα. Από το ΕΛΚ τον κύριο Μαλινό. Ευχαριστώ. Το θέμα βέβαια πονάει πολλές χώρες, όλους μας, αλλά κυρίως τις χώρες εκείνες που δυσανάλογα δέχονται αυτή τη τεράστια μεταναστευτική πίεση. Το κείμενο που έχει ετοιμάσει η συντάκτρια γνωμοδότηση το βρίσκω πολύ καλό, ισορροπημένο, οπότε τρία θέματα ουσίας, τρεις τροπολογίες έχω. Το ένα έχει να κάνει με το θέμα των αδικιών του συστήματος του Δουβλίνου. Όλο αυτό το έχετε συμπεριλάβει από ό,τι κατάλαβα. Κατά τα άλλα, για να μην μακρηγορήσω, θέλω να προσθέσω κάποια διευκρίνηση και επιμένω πρέπει να αποτελεί μέρος του προβληματισμού μας εφ' εξής. Αγωνιζόμαστε. Ζητάμε τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά μας σύνορα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Εμείς όμως πρέπει να βρούμε μια λύση που να πείθει όλους. Ναι, όλες οι κρίσεις είναι στη Μεσόγειο. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τα θαλάσσια μας σύνορα, δεν είναι μόνο αυτά που βρίσκονται υποποίηση, αλλά και τα χερσαία. Μπορεί να μην είναι πολύ δημοφιλές αυτό που λέω και πολλοί να μην το γνωρίζουν, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και στα χερσαία σύνορα μεταξύ της Βουλγαρίας και της Τουρκίας για παράδειγμα. Είμαι από τη Βουλγαρία και δεν τη γνώριζα αυτή την πίεση πριν από λίγα χρόνια. Όμως νομίζω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το εξηγήσουμε. Οπότε ή να μιλήσουμε εδώ για εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παριθμίσουμε τις χώρες ή να λέμε θαλάσσια και χερσαία σύνορα. Και να είμαστε σαφείς από αυτού. Έχουμε και χερσαία σύνορα τα οποία πρόκειται να είναι ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία επειδή η Τουρκία δεν εφαρμόζει τη συμφωνία επανεισδοχής. Και εδώ είναι που έρχομαι στη δεύτερη πρότασή μου. Και επιμένω γιατί έχει να κάνει και με το μέλλον του ζητήματος αυτού. Θέλω να υπογραμμίσουμε ότι η εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής πρέπει να συζητιούνται ιδιαίτερα με τις υποψήφιες χώρες για, για, για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Τουρκίας έχει να κάνει με την Τουρκία βέβαια, αλλά και στο μέλλον πρέπει να αποτελεί ένα βασικό σημείο των συνομιλιών που γίνονται για διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις συμφωνίες μας με τις χώρες της υποψήφιες για ένταξη πρέπει να το συμπεριλαμβάνουμε. Θα ήταν καλό πιστεύω για το μέλλον να συμπεριληφθεί εδώ στο κείμενο κάτι τέτοιο για την ε, μελλοντική εφαρμογή οτιδήποτε αποφασίσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Από το ECR, ο κύριος Μαριάς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση περιέχει πάρα πολλά στοιχεία σημαντικά. Ήθελα λίγο να σταθώ σε δύο σημεία που έχουν σχέση ε, με τις τεράστιες πιέσεις πραγματικά που δέχονται τα κράτη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερθώ στην Ελλάδα και στην Ιταλία, αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο θαλάσσια τα σύνορα, είναι και χερσαία, όπως αναφέρθηκε ο συνάδελφος ε, από τη Βουλγαρία. Διότι δεχόμαστε πιέσεις τεράστιες. Και να εξηγήσω ότι ούτως ή άλλως στην Ελλάδα υπήρχαν χιλιάδες παράνομοι μετανάστες εδώ και πολλά χρόνια. Προσθέστε τώρα δύο ζητήματα σημαντικά. Πρώτον, τους χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται καθημερινά στην Ελλάδα, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, εκεί είναι μεγάλη πίεση και όχι τόσο στα χερσαία σύνορα, στον Εύρο. Να προσθέσετε την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με ανθρωπιστική κρίση και που η άσχημη αυτή οικονομική κατάσταση θα ενταθεί, θα γίνει χειρότερη μετά την επιβολή των νέων μέτρων που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χτες. Επομένως καταλαβαίνετε ότι οδηγούμαστε στην Ελλάδα κυρίως σε μια εκρηκτική κατάσταση. Είναι αδύνατον να αντέξει η πατρίδα μου αυτή την τεράστια πίεση που έχουμε με χιλιάδες πλέον πρόσφυγες. Δεν είναι αδύνατο να φιλοξενηθούν. Και τα ποσά που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ψίχουλα σε σχέση με, τα με την τεράστια αδυναμία που έχει η πατρίδα μου να φιλοξενήσει τους χιλιάδες πρόσφυγες. Προσθέστε σε αυτό ότι, η Τουρκία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της ε, σε σχέση με τις συμβάσεις επανεισδοχής και μάλιστα υπήρχε πριν λίγες μέρες ένα δημοσίευμα στη Χουριέτ που αποκάλυπτε ότι οι τουρκικές αρχές διευκολύνουν όλο αυτό το λαθρεμπόριο ανθρώπων, την παράνομη μετακίνηση προσφύγων κυρίως από τη Συρία προς την Ελλάδα. Επομένως θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να καταργηθεί το Δουβλίνο 2. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μια αποθήκη ψυχών. Χιλιάδες άνθρωποι είναι εκεί εγκλωβισμένοι. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει αυτή η ρήτρα κατανομής. Δηλαδή ανάλογα με τον πληθυσμό, την έκταση, το ΑΕΠ που έχει κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάλογα με το πόσο ανεργία έχει ή όχι πρέπει να γίνει αυτή η κατανομή των προσφύγων και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αυτό να αφορά και την παράνομη μετανάστευση όχι μόνο τους, ε, τους πρόσφυγες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην Ελλάδα θα έλεγα και συνολικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προβλήματα θα ενταθούν και τουλάχιστον ε, σε αυτό το σύντομο περιεχόμενο της ε, γνωμοδότησης, γιατί δεν μπορεί να είναι εκτεταμένη, φύγονται σημαντικά ζητήματα και αυτά που έβαλα νομίζω πρέπει να ληφθούν υπόψη για να μπορούμε να έχουμε μια σφαιρική ε, αντιμετώπιση όσο μπορούμε ως Επιτροπή Αναφορών στα θέματα αυτά και κατά τα άλλα συμφωνώ με την εισήγηση της, που έκανε η συνάδελφος για την γνωμοδότησή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Εύη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω την εργασία της συναδέλφου ε, στην οποία βρίσκω πολύ θετικά. Εγώ όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα ζητήματα. Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια παράλογη κατάσταση. Δηλαδή, ε, οι, οι διακινητές ε, στην ουσία ε, κινούνται σε, που, βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν την θαλάσσια διαδρομή κινούνται σε ένα νομοθετικό κοινό, κενό. Μία από τις λύσεις που ε, το κίνημα των πέντε αστέρων προτείνει είναι ε, η δημιουργία νομίμων, νομίμων οδών μετακίνηση των ανθρώπων αυτών έτσι ώστε να χτυπηθεί στη ρίζα όλο αυτό το κακό το οποίο προκαλεί τόσα θύματα ε, και κάνει τη Μεσόγειο στην ουσία νεκροταφείο. Ε, στα εξωτερικά σύνορα της ε, Ευρώπης ε, γιατί σε αυτές τις περιοχές η κατάσταση είναι, έχει φτάσει σε σημείο που δεν μπορεί να προχωρήσει πια και να συνεχίσει. Επομένως, να ανοίξουν νόμιμες οδοί με δημιουργία κέντρων, με αναγνώριση επιτόπου στις χώρες στις ε, γειτονικές ή σε χώρες ε, στις οποίες έχουμε συγκρούσεις ένοπλες, να δημιουργηθούν επομένως ε, μορφές στήριξης έτσι ώστε να στηριχτούν επιτόπου ε, οι άνθρωποι αυτοί. Δεύτερον, ε, εγώ είμαι Ιταλίδα, εκπροσωπώ την Ιταλία ε, σε αυτό το κοινοβούλιο και πραγματικά αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι θα πρέπει να ελεγχθούν συστηματικά τα κονδύλια τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει για, την, για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και για τη διαχείριση γενικά αυτού του προβλήματος, διότι επανειλημμένα έχουμε δει κακή χρήση αυτών των κονδυλίων και από την κακή χρήση ε, προκύπτουν ε, πολλές ε, καταστάσεις διαφθοράς, έλλειψης διαφάνειας, περιπτώσεις που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχουν και επομένως βάσει αυτών των προβληματισμών καταλαβαίνετε ότι στα πλαίσια μιας ε, μεγάλης ε, επίγουσας κατάστασης δημιουργούνται και άλλες επίγουσες καταστάσεις οι οποίες εν τέλει αποβαίνουν κατά των ε, μεταναστών. Έχουμε παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων που από τις οποίες προκύπτουν ότι περισσότερα χρήματα κερδίζει κανείς από την παράνομη διακίνηση μεταναστών από ότι από το εμπόριο ναρκωτικών. Επίσης έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για την κακή λειτουργία των κέντρων υποδοχής. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Ε, είναι γεγονός ότι μπορεί τα προβλήματα αυτά να έχουν πιο τοπική διάσταση, ωστόσο τα κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούνται είναι ευρωπαϊκά, προέρχονται από την Ένωση και επομένως είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Άρα χρειάζεται και μεγαλύτερη ε, προσοχή και περισσότερος έλεγχος. Από την άλλη πλευρά είναι το θέμα του κανονισμού του Δουβλίνου δεν είναι δυνατόν να εξακολουθήσουν αυτές οι χώρες της πρώτης ε, πρόσβασης των μεταναστών να εξακολουθούν σαΐ, να είναι υπεύθυνα, υπεύθυνες για τους μετανάστες. Θα επανέλθουμε όμως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βαλέρο από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πολλά πράγματα μέσα σε ένα σύντομο κείμενο, δύσκολο να βάλει, να βάλει ε, όλα αυτά που χρειάζονται σε ένα τόσο ε, σύντομο κείμενο. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικής ποιότητας το κείμενο που μας έχει υποβληθεί. θα πρέπει να έχουμε, λέμε, ολιστική προσέγγιση του θέματος της ε, Μεσογείου, αλλά τότε θα πρέπει να δούμε και ολόκληρο το φάσμα της ε, μετανάστευσης. Ε, ίσως εύκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι είναι πρόβλημα μόνο της Μεσογείου, αλλά όχι, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Επίσης, αυτός ο μηχανισμός μετεγκατάστασης. Νομίζω καλό θα ήταν να πούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και την επιλογή ε, του ε, πρόσφυγα ε, δηλαδή ε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη χώρα τους ίσως έχουν και κάποιες προσωπικές προτιμήσεις με την έννοια ότι ε, υπάρχει μεγαλύτερη κοινότητα της χώρας του σε μια συγκεκριμένη χώρα ή έχει συγγενείς κτλ. Πρέπει λοιπόν οι ατομικές επιλογές και προτιμήσεις να ληφθούν και αυτές υπόψη. και στο σημείο 9, υπό το 9 θα ήθελα ε, να πω κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπε η από την FDD. Καλό είναι να μιλήσουμε για τους λόγους ε, που ε, οδηγούν τους ανθρώπους αυτούς να μεταναστεύσουμε οποιοδήποτε τρόπο και ενδεχομένως να δημιουργήσουμε αυτά, αυτές, αυτούς τους νόμιμους διάβλους. Γιατί μπορούμε να λύσουμε ένα κομμάτι του προβλήματος ε, μέσα από τη δημιουργία νομίμων διάβλων μετανάστευσης είτε στη Μεσόγειο είτε και σε άλλα σύνορα γιατί διαφορετικά θα εξακολουθούμε να έχουμε μονάχα νεκρούς στα σύνορά μας. Ε, και ξέρω ότι για τους ε, πρόσφυγες βεβαίως υπάρχουν κάποιες τέτοιες νόμιμες διαδικασίες, αλλά εμείς λέμε ότι θα πρέπει και για τους μη πρόσφυγες, για τους οικονομικούς μετανάστες, ε, να προβληφθούν και κάποιες νόμιμες οδοί μετανάστευσης. Αυτά θα ήθελα, αυτά τα στοιχεία θα ήθελα να τα δω στην έκθεση. Η κυρία Αλβιών παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μίτση για την εργασία της και επειδή έχουμε λάβει πολλές αναφορές από πολίτες μας που ανησυχούν για τους θανάτους στη Μεσόγειο, για την πολιτική μας ασύλου, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Επιτροπή μας πρέπει να διατυπώσει επικρίσεις έναντι της πολιτικής μετανάστευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να αλλάξει εντελώ αυτή η πολιτική που κλείνει τα σύνορα, υψώνει τείχους, που τους βάζει σε κέντρα κράτησης, που σε πολλές χώρες ακολουθεί ρατσιστικές πρακτικές, που δεν σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις για το άσυλο και επιπλέον τους φορτώνει σε αεροπλάνα και τους επιστρέφει σε χώρες ε, και τους αφήνει στη μέση της ερήμου ορισμένες φορές. Ως Επιτροπή Αναφορών πρέπει να είμαστε η φωνή όλων αυτών που ζητούν η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της για τους θανάτους στη Μεσόγειο. Έχουμε διτή ευθύνη. Από τη μία έχουμε ευθύνη γιατί οι πολιτικές μας είναι αυτές που τους υποχρεώνουν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Οι πολιτικές μας ε, έκαναν πολέμους, ε, οι κυβερνήσεις τους εξακολουθούν να απολούν ε, εξοπλισμούς και όπλα και επίσης και οι πολιτικοί που ακολουθούν πολλές από τις επιχειρήσεις μας. Και αυτές είναι πολλές από τις αιτίε που οφείλονται για τα θέματα αυτά. Και επιπλέον έχουμε και αυτή την πολιτική κλεισίματος των σύνορων. Όχι μόνο τους διώχνουμε από τις χώρες τους, αλλά τους κλείνουμε και την πόρτα στα σύνορά μας. Άρα χρειάζεται να διακυβεύσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι πολίτες της Ένωσης έχουν συνέστημα αλληλεγγύης πολύ περισσότερο από τις κυβερνήσεις τους. Από τις κυβερνήσεις που έχουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να ακουστεί η φωνή της κοινωνίας των πολιτών που είμαι σίγουρη ότι αυτό που ζητάει είναι ότι κανείς δεν θα πρέπει να χρειαστεί να φύγει από τη χώρα του και αν είναι υποχρεωμένος να φύγει δεν θα πρέπει να παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα στην Μεσόγειο. Γι' αυτό πρέπει να ζητήσουμε νόμιμες δυνατότητες μετανάστευσης. Πρέπει να μπορεί να ζητούν διεθνή προστασία στις πρεσβείες, να βελτιώσουμε την επανένωση των οικογενειών και το σύστημα ασύλου. Πρέπει λοιπόν να επικρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι Θέλει περισσότερη Frontex, περισσότερη στρατιωτικοποίηση της Μεσόγειο, περισσότερη εξωτερικοποίηση των συνόρων. Όλα αυτά δεν είναι λύσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να καταστεί σαφές ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η επιχειρηματολογία προστασίας των συνόρων, γιατί δεν υπάρχει εχθρός για να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για προστασία και άμυνα στα σύνορα και πραγματικά είναι θλιβερό αυτό που ακούω, ορισμένοι λένε ότι ανησυχούν περισσότερο για την πίεση που υφίστανται οι χώρες τους από το ότι έρχονται μετανάστες και πρόσφυγες και όχι για τη ζωή αυτών των ατόμων. Εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Αριστερά, θα συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, στη γνωμοδότηση και όπως σας είπα θα μεταφέρουμε τις ανησυχίες που οι πολίτες μας αναφέρουν. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και πρόεδρος. Είμαι σκιώδης της Άλντε για το θέμα αυτό. Πρώτα λοιπόν και εγώ να ευχαριστήσω την συντάκτρια, την κυρία Μίτση. Η γνωμοδότηση αυτή νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη για να συμβάλλουμε στην εντολή που δόθηκε από την Ολομέλεια στη Λίμπε για να υπάρξει μια σφαιρική, μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος. Η συμβολή της Επιτροπής μας σε αυτήν την ευρή έκθεση βασίζεται στις αναφορές που έχουμε λάβει. Έχουμε λάβει πολλές. Ορισμένες είναι από πολίτες της Ένωσης αναφέρονται σε πολλά θέματα που σχετίζονται με την κρίση της μετανάστευσης, εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για την ε, απώλεια ανθρωπίνων ζώων στη Μεσόγειο και για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το αντιμετώπισε με ευρωπαϊκό τρόπο. Είναι θέμα κατανομής ευθύνης, είναι θέμα δράσης από κοινού της Ένωσης και στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης λοιπόν είτε είναι χερσαία είτε θαλάσσια. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία μαζί σας να μην πάρω περισσότερο χρόνο. Θα συνεργαστούμε. Ο κύριος Άκερ τώρα. Ευχαριστώ. Δεν αντιμετωπίζει τους λόγους για τους οποίους προσελκύονται τα άτομα στην Ένωση. Είναι μια κρίση που ξεκινάει στη Μεσόγειο φτάνει μέχρι το Καλέ και έχουμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο 325.000 κάθε χρόνο καθαρή μετανάστευση έχουμε. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στις ιατρικές υπηρεσίες. Φτάνει, φτάνει πια. Στην ουσία τώρα δρέπουμε τους καρπούς από την καταστροφική πολιτική που ακολουθήσαμε εδώ και 10-15 χρόνια. Βομβαρδίσαμε τη Μέση Ανατολή και προσπαθούσαμε να επιβάλλουμε τη δημοκρατία με τα όπλα. Και τώρα έχουμε αφήσει εκεί κατεστραμμένα κράτη. Γι' αυτό έχουμε αυτή την κρίση. Αλλά γιατί έρχονται. Γιατί δεν αντιμετωπίζουμε τους λόγους που τους προσελκύουν. Το πρώτο είναι η ελεύθερη διακίνηση. Έρχονται εδώ, εξοπλούν το Σέγγεν και περνάνε από το ένα κράτος της Ένωσης στο άλλο. Γι' αυτό στο καλέ βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Όλη αυτή η παράτητη μετανάστευση μετανάστες κινδυνεύουν τη ζωή τους, σκαρφαλώνουν σε τρένα για να μπουν στον Αμένο Βασίλειο. Γιατί να μην πάρουμε μαθήματα από την Αυστραλία, πώς αντιμετωπίζει η Αυστραλία όλα αυτά τα καράβια του μετανάστες. Η Αυστραλία έχει ε, προσέγγιση μηδενικής ανοχής. Αντιστρέφουν τη ρότα των πλοίων και έτσι σταμάτησε να προσελκύει η Αυστραλία μετανάστες. Αντί λοιπόν να προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο κατανομής των μεταναστών σε όλες τις χώρε της Ένωσης, θα έπρεπε να πούμε φτάνει. Να χτυπήσουμε το πόδι μας στο έδαφο. Δεν θα είναι όλα ανοιχτά για όλους. Θα τα σπρώξουμε τα καράβια, θα τα αναγκάσουμε να αλλάξουν πορεία. Η συζήτηση για τη μετανάστευση βέβαια στη χώρα μου γίνεται εδώ και χρόνια. Και επιτέλους έγινε αποδεκτό ως θέμα για δημόσια συζήτηση το θέμα της μετανάστευσης για την νόμιμη μετανάστευση. Αυτό που προσελκύει πολύ στον ΕΒ Βασίλειο είναι το σύστημα επιδομάτων που έχουμε και παροχών. Η κυβέρνηση έχει σχέδια ότι μόνο από τρει μήνε και αν κερδίζει 155 λίρε τη βδομάδα θα δικαιούνται επιδομάτων εργασία. Το σύστημα παροχών τώρα που έχουμε, ένα ένας ε, ε, γονιός που μεγαλώνει μόνο του δύο παιδιά και δουλεύει 16 ώρες τη βδομάδα, λαμβάνει 116 για επίδομα παιδιών, 144 στεγαστικό απείρωμα και 34 άλλο επίδομα παιδιών. Οπότε το εβδομαδιαίο εισόδημά τους ανεβαίνει στις 500 λίρες. Και από, αυτά τα 500, από αυτές τις 500 λίρες κερδίζει μόνο 155. Οπότε ετησίως κερδίζει 8.000 από την εργασία του και 12.000 από τα επιδόματα. Αυτό δημιουργεί τρομερό πρόβλημα στο φορολογικό μας σύστημα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ε, συνεχίσει να ισχύει αυτό το σύστημα και το δικό μου το κόμμα λέει ότι πρέπει για πέντε χρόνια να εργάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο πριν να αποκτήσει δικαίωμα σε αυτέ τι παροχέ. Λοιπόν, θα φωτοτυπήσω αυτό το κείμενο και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό για μένα, γιατί το κείμενο αυτό και για το κόμμα μου, γιατί το κείμενο αυτό λέει ότι δεν μπορούμε να μην εφαρμόσουμε του κανόνε ελεύθερη διακίνηση. Δεν έχει καμία δυνατότητα η Βρετανία να μπορέσει να προστατεύσει τα σύνορά τη, αλλά δεν έχει καμία δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν θα γίνει το δημοψήφισμα, γιατί αυτό το θέμα θα παίξει ρόλο στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο Πρόεδρο. Εντάξει, είναι δικό σα θέμα αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και δεν έχουμε αναφορές για το θέμα αυτό. Η κυρία Μίτσι κάνει θαυμάσια δουλειά, συντάσσοντας την αναφορά, με βάση, συγγνώμη, συντάσσοντας τη με βάση τις αναφορές που έχει λάβει η Επιτροπή μας. Σε άλλες επιτροπές μπορεί από άλλη άποψη να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση. Εδώ βασιζόμαστε στις αναφορές που έχουμε λάβει. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα τώρα. Προθεσμία για τροπολογίε 22 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 17 Σεπτεμβρίου. Στη Λίμπε 16 Νοεμβρίου το αργότερο. Μπορεί να είναι και νωρίτερα. Αυτά. Να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Κυρία Αλμπιόλ, μα πήρατε το λόγο. Θέλετε να ξαναμιλήσετε γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο. Έχουμε κάποια καθυστέρηση. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Θέλω να πω ότι τίποτα από αυτά τα οποία ζήτησε η ομάδα μας στην Επιτροπή μας δεν έχει συμπεριλάβει η κυρία Μίτση από αυτά που έχει ζητήσει το UKIP. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμπεριλάβει η κυρία Μίτση. Δεν είναι δυνατόν να το λέμε αυτό για παιδιά τα οποία φεύγουν από ριωγμένη εξαιτία του πολέμου και άλλων βάρβαρων πράξεων. Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Ωραία. Προχωράμε στο σημείο 18. 59 του 12. Διακρίσεις σε βάρος υπηκών που δεν είναι μαλτέζικης υπηκότητας, ευρωπαϊκής υπηκότητας στη Μαλτά. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή, ο κύριος Λαβάτζη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω πραγματικά να αναφερθώ σε αυτό που εξετάζουμε τώρα. Είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2012, όπου είχαμε από τον αναφέροντα την αναφορά του. Και βάσει αυτής της αναφοράς ξεκινήσαμε ένα pilot και στείλαμε στις αρμόδιες χώρες μέλη τις ερωτήσεις μας. Ζητήσαμε Επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους είχε πρόβλημα ο αναφέρον από την Go PLC και την Μελίτα δηλαδή τους στείλαμε ερωτήσει και πήραμε τις απαντήσεις τους που λένε ότι η πρακτική αυτή του να ζητάει η εταιρεία εγγυήσεις έχει να κάνει με τους πελάτες οι οποίοι δεν είχαν ε, μαλτέζικη ταυτότητα. Βάσει όμως τις οδηγίες για τις υπηρεσίες και βάσει του άρθρου 20 σημείο 2 εξετάσαμε τις απαντήσεις των εταιριών και διαπιστώσαμε ότι τέτοιοι περιορισμοί για αγγίσεις, δηλαδή πριν υπάρξει σύμβαση, είναι κάτι το οποίο αιτιολογείται. Βάσει του ότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος, αν έχει δηλαδή κανείς ε, ταυτότητα Μάλτας, είναι ο μόνος τρόπος για να καταλάβει αν είναι αξιόπιστος ή όχι ο πελάτης. Και μετά από τρεις μήνες μπορεί να ζητήσει ταυτότητα Μάλτας κάθε διαφερόμενος, οπότε οι συνθήκες των συμβολέων λένε ότι άπαξ και κάποιος έχει την ταυτότητα αυτή μετά από τρεις μήνες που μένει στη χώρα, τότε η εγγύηση επιστρέφεται. Γι' αυτό λοιπόν και βάσει αυτής της αιτιολόγησης αποφασίσαμε το 2014 να κλείσουμε την υπόθεση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα, η κυρία Μίτση είναι η πρώτη. Ευχαριστώ. Σωστά τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν δύο μεγάλοι πάροχοι. Και ένας από αυτούς αμφισβητεί την καταγγελία. Γιατί δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε πολίτες εμείς της Μάλτας. Και άλλος πάροχος είπε ότι οποιαδήποτε εγγύηση ζητάτε επειδή δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Μάλτας κάποιος, όταν αλλάξουν οι προϋποθέσεις και είναι μόνιμος κάτοικος, παίρνει πίσω την εγγύηση. Γι' αυτό και έκλεισε η αναφορά αυτή. Ωραία, άλλος κανείς. Παρακαλώ κύριε Αντάλη. Μας έδωσε επιπλέον πληροφορίες ο αναφέρον, έχουμε αντίγραφα. και τότε όμως τα επιχειρήματα, για μένα το θέμα είναι περισσότερο ε, θέμα γιατί υπάρχουν αυτές οι απαιτήσει από μία επιχείρηση παρά το κατά πόσο γίνεται διάκριση ανάμεσα σε Μαλτέζους ή άλλους Ευρωπαίους πολίτες που δεν είναι όμως Μαλτέζοι. Οπότε, Ακόμα και αν λάβουμε υπόψη μας τα διάφορα επιχειρήματα, κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες ή δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες για να καταλάβουμε κατά πόσο υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε Μαλτέζους και μη Μαλτέζους. Ακόμα και αν υπάρχουν οι επεξηγήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά δεν αναφέρεται κάτι για το θέμα της υπηκότητας όπως ήταν η αρχική καταγγελία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η θέση του ΕΛΚ είναι επίσης να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Ωραία, καλώς. Κανένας άλλος. Κατάλαβα ότι τα τέλη που πληρώνονται επιστρέφονται μετά, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος. Αυτό ισχύει, έτσι. Ωραία. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι θέλουμε να κλείσουμε την ε, αναφορά. Καλώς. Συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι κάτι αντίστοιχο. Φίλια ε, του 2013, πάλι πρόκειται για διακρίσεις στη Μάλτα, σε σχέση με ηλεκτρονική κατοικία. Δεν είναι ούτε και αυτός αναφέρον εδώ, γι' αυτό και δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Λιού, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο έχει λάβει ήδη δύο ε, αναφορές σχετικά με την ε, διαδικασία ε, της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής στην Μάλτα για περιπτώσεις ε, εγγράφων που έχουν εκδοθεί μετά την, ε, συγγνώμη, πριν ε, από τον Ιανουάριο του 2013. Οι αρχές της Μάλτας άλλαξαν άλλαξαν την μορφή των εγγράφων και πλέον δίνουν μία πλαστική κάρτα παραμονής ε, και από εκεί προέκυψαν τα προβλήματα. Ξέχασα να σας πω προηγουμένως ότι αυτή η διαδικασία ε, απολύτως ευθυγραμμίζεται <clears throat> με την ελεύθερη κυκλοφορία στο, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και να σας πω επίσης ότι οποιοδήποτε εγκαθίσταται στην Μάλτα μετά από τρεις μήνες μπορεί να ε, ζητήσει την ε, άδεια παραμονής στην χώρα αυτή. Ήρθαμε σε επαφή με τις αρχές της Μάλτας οι οποίες διευκρίνησαν ότι η διαδικασία για να πάρει κανείς αυτήν τη νέα σε πλαστική μορφή κάρτα Ε, χρειάζεται απλώς να δώσουν οι πολίτες τα, την έγγραφη μορφή, δηλαδή αυτά τα ε, έγγραφα τα οποία έχουν σε χάρτινη μορφή, ε, έτσι ώστε να τους δοθεί η, η κάρτα. Μπορούν επίσης με το ταχυδρομείο να κάνουν τη διαδικασία αυτή. Μέσω της ε, κάρτας αυτής μπορούν λοιπόν να κυκλοφορήσουν, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας κτλ. Ε, After another contact in August 2013, τον Αύγουστο του 2013 οι αρχές της ε, Μάλτας αναγνώρισαν ότι είχαν προκύψει καθυστερήσεις στην αποστολή των πλαστικών καρτών ε, και ότι αυτό οφείλεται σε περιορισμένους διοικητικούς ε, πόρους. Ε, ωστόσο είπαν ότι υπήρχε συγκεκριμένη πρόθεση αύξησης των υπαλλήλων που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Ε, η Κομισιόν ε, θεωρεί ότι έχει πλέον ε, ομαλοποιηθεί η κατάσταση, άλλωστε δεν έχει ληφθεί και κάποια επιπλέον αναφορά όσον αφορά αυτήν την πλαστική μορφή της άδεια παραμονής ή της ταυτότητας. Η κυρία κυρια Μίτσι, να σας επιβεβαιώσω ότι οι αρχές της Μάλτας όντως δίνουν πλέον μία νέα ταυτότητα ε, η οποία περιλαμβάνει και ε, στοιχεία για την ε, ασφάλεια και τα λοιπά και που αφορά τους μη υπηκόους Μάλτας, δηλαδή υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όχι της Μάλτας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον οποιοδήποτε πρόβλημα και ε, δεν υπάρχει καμία παραβίαση των συνθήκων από πλευράς της ε, ε, Μάλτας, γιατί άλλωστε το ίδιο ηλεκτρονικό έγγραφο έχουν όλοι οι πολίτες. Πρόεδρος, ναι, όντως ε, είχαμε την ε, αναφορά 0100 του David Rally, αλλά έχουμε και την 1419 του 13 ε, από πλευράς Φιλανδού ετούντος πάλι για, αυτήν, για αυτό το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης. Από ό,τι καταλαβαίνω όσον αφορά την πρώτη αναφορά, την κλείνουμε. Όσον αφορά τη δεύτερη, τι θέλετε να κάνουμε, αυτή του Φιλανδού υπηκόου. Είναι για το ίδιο θέμα, λέει η κυρία Μίτση. Ναι, ε, αφορά και τις ηλεκτρονικές κάρτες ε, αλλά και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού και νερού. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια περίπτωση. Ωραία, επομένως θέλετε να κλείσουμε και την 14-19. Ε, Πολύ ωραία, αυτό θα κάνουμε. Υπάρχει όμως και η αναφορά 10-12-2012, δηλαδή του 2013, ε, πάλι για διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τις, ε, ε, το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στη Μάλτα και στο νησί του Γκόθο. Σχετικά με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης ε, των ε, μη μαλτέζων υπηκών και έχουμε επίσης ε, και άλλη μία αναφορά σχετικά με εξαιρετικά υψηλούς λογαριασμούς για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Θα δώσω ξανά τον λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα εδώ για τον ηλεκτρισμό και την ίδρυυση. Το πρώτο ήταν ε, διαφορετικές ε, τιμές για πολίτες από άλλες χώρες. Αυτό αφορούσε και την 14-19. Και την 10-12 του 13. Η νομοθεσία στη Μάλτα προβλέπει τρεις διαφορετικές τιμές για τον οικοκυριό, για αυτούς που διαμένουν και αυτούς που δεν διαμένουν. Έχουμε λάβει 15 διαμαρτυρίες για τα θέματα αυτά, γιατί μη Μαλτέζοι πολίτες έπρεπε να πληρώσουν 30% παραπάνω. γιατί δεν είχαν αυτόματα δικαίωμα να λαμβάνουν τις, ε, να πληρώνουν τιμές ε, ανθρώπων που παραμένουν έπρεπε πρώτα να κάνουν κάποιες διοικητικές διαδικασίες να πάρουν ε, άδεια παραμονής ενώ οι Μαλτέζοι δεν χρειαζόταν να τα κάνουν αυτά ήταν αυτόματο και επειδή δεν θεωρούν το κάτοικοι στη Μάλτα δεν μπορούσαν να λάβουν κάποιες επιδοτήσεις κάποιο, κάποια μείωση για οικολογικούς λόγους και άλλα τέτοια. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ήρθαμε σε επαφή με τις αρχές της Μάλτας και χρειάστηκε να κάνουμε συζητήσεις ανοιχτά και ξεκινήσαμε η διαδικασία επί παραβάση τον ε, Δεκέμβριο του 2012 γιατί η απάντηση που λάβαμε δεν ήταν ικανοποιητική. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία επί παραβάση άλλαξαν το 2014 οι αρχές της Μάλτας στη διαδικασία υποβολής αίτησης και τώρα μπορούν να πάρουν τις φθηνότερες τιμές και οι άλλοι κάτοικοι κρατών μελών απλώς υποβάλλοντας μια αίτηση με ταυτότητα ή δελτίο ταυτότητας. Οπότε η Κομισιόν Επιτροπή, η Κομισιόν θεωρεί, συγγνώμη, ότι δεν υπάρχει θέμα διακριτικής μεταχείρισης πλέον και ζητήσαμε η Μάλτα να ξεκινήσει και μία διαδικασία για να επιστρέψει τα χρήματα σε αυτούς ε, που πλήρωσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα περισσότερα. Και αυτή η διαδικασία άρχισε να ισχύει τον περασμένο Μάιο. Ή μάλλον καλύτερα. Πρέπει να πω ότι μέχρι το Μάιο είχαν λάβει μόνο 43 αιτήματα για επιστροφή ε, τμήματος του λογαριασμού. Κάτι άλλο τώρα που αφορά ενίκους που έχουν ε, νοικιάσει σπίτια από Μαλτέζους ιδιοκτήτες. Για να πάρουν αυτά τα ωφελήματα πρέπει να υποβάλουν ε, μία αίτηση που πρέπει να έχει υπογράψει ο ιδιοκτήτη. Και αν δεν υπογράψει ο ιδιοκτήτη, δεν μπορούν να έχουν αυτή την καλύτερη τιμή. Όλα αυτά τα αναφέρει η αναφορά 1737 του 13. Και νομίζουμε ότι μπορεί να ισχύει και το 1655 του 14, αλλά δεν είναι πολύ συγκεκριμένη. Απλώς λέω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα για τους κατοίκους, για τους πολίτες άλλων ε, κρατών μελών. Δεν ξέρουμε αν είναι για τους ε, ενοικιαστές. Δεν είναι σαφής αυτή η αναφορά. Για το θέμα αυτό ήρθαμε σε επαφή τον Νοέμβριο του 2014 με την Μάλτα. Έχουμε κάνει διάφορες συναντήσεις έκτοτε. Η τελευταία έγινε 24 Ιουνίου πριν από λίγες εβδομάδες. Μέχρι στιγμής η απάντηση των αρχών της Μάλτας δεν είναι ικανοποιητική. Λένε ότι οι οργανισμοί κοινή ωφέλεια δεν μπορούν να ξέρουν τι γίνεται. Το συζητάμε όμως ακόμη. Περιμένουμε και άλλες απαντήσεις μετά αυτή τη συνάντηση τον Ιούνιο. Το θέμα αυτό σαφώς ακόμη δεν έχει επιληθεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς που θέλει τον λόγο η μαρλενα Ναι, όπως είπαμε υπάρχουν διαφορετικά τιμολόγια, όπως είπε η επιτροπη Αλλά πολλά από αυτά τα διαφορετικά τιμολόγια έχουν ε, καταργηθεί. Και η πάροχη υπηρεσιών Unlimited Limited έχει έναν ε, μηχανισμό για την αντιμετώπιση των παραπώνων. Όποιος έχει να κάνει ένα παράπονο, βλέπει κάποιον υπάλληλο της εταιρεία και αποζημιώνεται και συχνά. Δεν είναι τόσο σαφής η κατάσταση όπως θα θέλαμε, αλλά πολλά από τα προηγούμενα προβλήματα, πριν από τον Ιούλιο του 2013 δηλαδή, έχουν επιληθεί. Λόγω και αυτού του μηχανισμού επανόρθωσης. Η κυρία Ντάλη, αν κατάλαβα καλά, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα. Και από ό,τι κατάλαβα λοιπόν η Κομισιόν λέει ότι δεν υπάρχουν διαφορετικά τιμολόγια για Μαλτέζους και μη. Αλλά δεν θεωρεί ότι οι υπηρεσίες κοινή ωφέλεια τιμολογεί τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή. και αν ο λογαριασμός πάει στον ε, ενοικιαστή πληρώνει περισσότερα. Κοιτάξτε. Το τιμολόγιο για τους κατοίκους δίνονται για όσους έχουν την πρώτη τους κατοικία στην Μάλτα και όσοι έχουν ένα γκαράζ ή ένα εξωτικό σπίτι πληρώνει με άλλο τιμολόγιο Αλλά το πρόβλημα που προκύπτει είναι αν υπάρχει θέμα μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Αυτό έχει θέσει μια συγκεκριμένη αναφορά. Δεν βλέπω εδώ καμία διακριτική μεταχείριση μεταξύ Μαλτέζων ή όχι κατοίκων της Ένωσης. Εάν η υπηρεσία κοινή ωφέλεια βασίζεται στο κριτήριο εάν ο λογαριασμός αφορά μια πρώτη ή δεύτερη κατοικία. Όποιος νοικιάζει θα πληρώσει περισσότερο. Επειδή υπάρχει αυτό το θέμα με τον ιδιοκτήτη. Αλλά πώς είναι δυνατόν ε, ένας οργανισμός ηλεκτρισμού ίδρυυσης να έχει την ευθύνη να διευκρινίσει μια διαφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή Εάν δηλαδή θα δώσει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή να εκδώσει το λογαριασμό στο όνομά του ή όχι. Μισό λεπτό, είναι και άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Ο κύριος Πάρα. Η θέση του κόμματός μας είναι ότι έχουμε τρεις αναφορές εδώ για την πρώτη 10-12 φαίνεται ότι έχει επιληθεί το θέμα αυτό άρα καλό θα ήταν να την κλείσουμε για τις δύο άλλες 17-37 και 16-55 βλέπουμε ότι ότι δεν είναι απόλυτα σαφής η κατάσταση Άρα να περιμένουμε για τις επόμενες συζητήσεις ε, Επιτροπής Μάλτας. Οπότε καλύτερα να τις κρατήσουμε ανοιχτές. Αυτή είναι η θέση μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Θέλει να προσθέσει τίποτα η Επιτροπή ή μπορούμε να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Βεβαίως να απαντήσετε, να απαντήσετε. Για τις διακρίσεις για τους ενοικιαστές. Δεν είναι άμεση διάκριση αλλά είναι έμεση, σαφώς, διότι ξέρουν τις διαφορετικές ε, τιμές όσοι μένουν στη Μάλτα. Ένας πολίτης της Ένωσης φτάνοντας στη Μάλτα μπορεί να μην έχει πληροφόρηση. Και πληρώνει περισσότερα. Είναι πρόβλημα λοιπόν που κυρίως αντιμετωπίζουν στην πράξη οι μη Μαλτέζοι. Η ε, κυρία Ντάλη. Μα εγώ κατάλαβα ότι είναι θέμα για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλης να ενημερώσουν τους ε, καταναλωτές πρόεδρος. Αν κατάλαβα και εγώ, προτείνεται να κλείσουμε τη 10-12 και συμφωνεί και η Επιτροπή γιατί δεν έχει αντίρρηση. Για τη 16.55 και τη 17.37 προτείνω να μείνουν ανοιχτές και να ζητήσουμε γραπτή απάντηση από την Επιτροπή και να στείλουμε ένα γράμμα και στην ε, μόνιμη αντιπροσωπεία της Μάλτας να τους θέσουμε τα θέματα που θέτουν οι αναφορές και όταν πάρουμε μια εμπεριστατωμένη απάντηση τότε να δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Καλώς, το επόμενο θέμα. Θέμα 21 στην ημερήσια διάταξη. Ακούστε. 1098 του 2010 ενό γερμανική ηθαγένεια πολίτη σχετικά με διακρίσει ει βάρο πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τι ειδικέ Αρχέ. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Ενώ σου προεδρεύω τη Επιτροπή Αυτή και υπάρχει και άλλη μια αναφορά, η 1183 του 2010 πάλι Γερμανού πολίτη, σχετικά με την αναγκαιότητα ενό προσωπικού αριθμού μητρώου στη Σουηδία. Και υπάρχει και μια τρίτη, η 1289 του 2012, Βρετανού υπηκόου, για παραβίαση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία και κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σουηδική Μόνιμη Αντιπροσωπεία έχει προσκληθεί, αλλά είπε ότι δεν θα έρθει. Δεν είναι εδώ ούτε αναφέροντες, οπότε θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα έχουμε πάλι την κυρία Λου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Οι αναφορές αυτές έχουν να κάνουν με πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι δεν καταφέρουν να έχουν ένα νούμερο καταχώρησης σε μετρό στη Σουηδία. Και αυτό γιατί δεν ήταν κάτι και πάνω από έξι μήνες στη Σουηδία. Και σε μία περίπτωση πρόκειται για πιο προσωρινή διαμονή. Αν δεν έχεις αυτόν τον αριθμό μητρώου, η ζωή σου γίνεται πολύ δύσκολη στη Σουηδία από ό,τι φαίνεται. Η προϋπόθεση για να πάρει κανείς αυτό το προσωπικό αριθμό ταυτότητας είναι να πρέπει προηγουμένως να έχεις γραφτεί στα Σουηδικά Μητρώα Πληθυσμού. Σύμφωνα με τη Σουηδία, τα... οι πολίτες δεν μπορούν να καταγραφούν στα Μητρώα αυτά πληθυσμού αν δεν μπορούν να αποδείξουν ότι κατοικούν στη Σουηδία πάνω από ένα χρόνο και όταν κάποιος δεν τηρεί τις προϋποθέσεις αυτές έχει έναν, ένα νούμερο συντονιστικό το οποίο όμως δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο όπως σαν να είχε τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας. Όταν άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να ερευνά το θέμα αυτό, διαπιστώσαμε ότι το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν διάφοροι Ευρωπαίοι πολίτες. Γιατί μπορεί κανείς να πάει για λιγότερο από ένα χρόνο ως φοιτητή ή για προσωρινή απασχόληση για οτιδήποτε σε μια άλλη χώρα. Η προπόθεση αυτή του ενός έτους κατοικίας επιβάλλεται σε οποιονδήποτε ζητάει τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας. Οπότε είτε εργαζόμενοι, είτε αυτοπασχολούμενοι, είτε φοιτητές, καταναλωτές, οτιδήποτε ή τα μέλη της οικογένειας τέτοιων ατόμων ε, χρειάζονται αυτόν τον ε, αριθμό και δεν μπορούν να τον έχουν. Ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας επίσης είναι αναγκαίος και για οποιαδήποτε επαφή με τις διοικητικές αρχές της Σουηδίας αλλά και για τις επαφές με ιδιωτικές υπηρεσίες για να έχει σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου οι τράπεζες επίσης για να ανοίξει κανείς λογαριασμό τραπεζικό χρειάζονται αυτόν τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας. Και αυτό που είναι ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι χρειάζεται κανείς αυτόν τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας, το PIN όπως το λένε, για να μπορέσει να έχει επαφή διαδικτυακά με τη Σουηδική δίκη. Δεν μπορεί να μπει μέσα, να κάνει login αν δεν έχει αυτό το νούμερο. Και το χειρότερο για μας είναι ότι δεν μπορείς να έχεις περίθαλψη χωρίς αυτόν τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας. Πας δηλαδή εγκαθίστασαι στη Σουηδία, δεν έχεις πια εκάλυψη ασφαλιστική από τη δικιά σου τη χώρα, η Σουηδία όμως δεν σου επιτρέπει να επωφεληθείς από το δικό του σύστημα γιατί σου δίνει αυτόν τον αριθμό. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο, βάσει της οδηγίας 2004-38, τίθενται τα κριτήρια πώς μπορεί κάποιος νόμιμα να κατοικεί σε μια άλλη χώρα. Και λέμε ότι πρέπει να έχει κάποια οικονομική δραστηριότητα ή να έχει επαρκείς πόρους ή πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. δεν υπάρχουν ε, άλλες προϋποθέσεις που να μπορούν να επιβληθούν. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε επαφές με τις ειδικές αρχές όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2004-38 για την ελεύθερη διακίνηση. Ξεκίνησε η διαδικασία επί την παραβάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των Σουδικών Αρχών. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ακόμα και με άλλες επαφές που είχαμε από την Γενική Διευθύνση Απασχόλησης και τον ίδιο τον Επίτροπο, οι Συνδικές αρχές πρότισαν υποσχέθηκαν ότι θα διευθετήσουν το θέμα και θα υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις προς λύση. Καλώς, ναι. Βάλτε με τι ειδικέ αρχέ Πίτερ, γιατί πραγματικά είναι απίστευτο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιο στη Σουηδία ούτε μισή μέρα χωρί να έχει αυτόν τον ε, προσωπικό αριθμό ταυτότητα. Το ξέρω. Οπότε ναι, προτείνω λοιπόν τα εξή. Πρώτον, αν μπορούμε να στείλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή μια πολύ αυστηρή απάντηση, όταν την έχουμε, μέσα σε μερικές μέρες δηλαδή, τότε εμείς θα στείλουμε επιστολή τις αρχές ειδικέ εδώ στις Βρυξέλλες, θα ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες και θα επιμείνουμε ότι αν δεν γίνει τίποτα από τι ειδικέ αρχές, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ερευνά, προσπαθεί να δει αν μπορεί να υπάρξει κάποια λύση, αλλιώ θα υπάρξει πάλι διαδικασία επί την παραβάση κατά της Σουηδίας. Καλό θα κάνει, θα είναι η πρώτη φορά. Ποτέ δεν έχει γίνει. Θα ήταν πολύ χρήσιμο. Συμφωνείτε? Ναι, Πίτερ, Συμφωνεί. Καλώ. Τώρα έχουμε ένα θέμα ακόμα στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Πάντα μαχίζει κανείς στι 9 και έχει φτάσει 6 και, δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, επόμενο θέμα είναι η αναφορά 0026 του 2012 για διακρίσεις βάσει του φύλου Ιταλία και η άλλη το 2012, επίσης που έχει να κάνει με την ηλικία συνταξιοδότηση στην Ιταλία. Δεν είναι εδώ οι αναφέροντες. Το λόγο έχει ο Αλβάρο Λιβέιρα ή κάσα Κόρονεν. Ποιος από τους δύο. Ευχαριστώ. Αλβάρο Λιβέιρα ονομάζομαι, πράγματι, και είμαι εδώ με τον συνάδελφο. Δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα θέματα εδώ και αρκετό καιρό και θέλω να σας ενημερώσω για το ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση. Οι υποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν με την νομοθεσία του 214 του Δεκεμβρίου του 2011 που αναφέρεται στις συνταξιοδοτήσεις και αναφέρονται λένε ότι υπάρχει μια διάκριση βάση φύλου σε βάρος των εργαζομένων ασθενικού φύλου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά θέλω να σας εξηγήσω λίγο το πλαίσιο. Όσον αφορά την πρόορη συνταξιοδότηση, υπάρχουν διαφορετικές προϋποθέσεις για τους άντρες και για τις γυναίκες. Εξαρτάται από τον αριθμό ετών συνεισφορά του εργαζόμενου προκειμένου να πάρει πρόορη σύνταξη. Με δύο λόγια, ένα χρόνο λιγότερο απαιτούν οι αρχές για πρόορη συνταξιοδότηση. Πώς έχει η κατάσταση σήμερα. Μετά από επαφές που είχαμε με τις Ιταλικές Αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πρόβλημα και έστειλε ε, μια επίσημη προειδοποίηση στις Ιταλικές Αρχές τον Οκτώβριο του 2013 με την οποία έλεγαν ότι υπάρχει παράβαση της 264 που έχει να κάνει με τις διακρίσεις στην απασχόληση. Πήραμε μια απάντηση τον Ιανουάριο του 2014 από τις Ιταλικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα αναλύει τις απαντήσεις των Ιταλικών Αρχών. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι πρέπει να κάνει. Θα με ρωτήσετε γιατί. Ε, θα σας πω ότι το θέμα είναι περίπλοκο. Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η υπόθεσή μας στην επιστολή που στείλαμε ήταν ότι η Ιταλική νομοθεσία παραβιάζει την αρχή της ισότητας όσον αφορά τα σταξιδοτικά δικαιώματα. Και για να το πω απλά, σημαίνει ότι δεν μιλάμε για τους νόμους που έχουν να κάνουν με ολόκληρη την κοινωνική ασφάλιση που εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά μόνο για ορισμένες κατηγορίες, όπως είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η Ιταλία όμως απάντησε ότι κατά τη γνώμη της δεν ισχύει αυτό. Κατά τη γνώμη της Ιταλίας, τα αξιωτικά δικαιώματα αφορούν όλους τους εργαζόμενους. Είναι καταστατικό δηλαδή συνταξιδοτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτεται από άλλη οδηγία, την 79-7, που έχει να κάνει με τα γενικά θέματα κοινωνικής ασφάλισης, που βάζει κάποιες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, για την ηλικία της εξεδότησης. Γι' αυτό λέω ότι είναι περίπλοκο το θέμα. Η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει αλλάξει ακόμα. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε νέα θέση αναθεώρησης, η αλλαγή της προηγούμενης θέσης μας, ούτε έχουμε αποφασίσει ότι θα μείνουμε σε αυτή. Αναλύουμε την υπόθεση ακόμα. Σας ευχαριστώ. Επιθυμεί κάποιος να λάβει το λόγο. Η Ελεονόρα. Παρακαλώ, Ελεονόρα, έχεις το λόγο. Στην πραγματικότητα, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό ε, το θέμα αυτό, αυτή η αναφορά, γιατί δεν έχουμε και πολλά καινούργια στοιχεία. Πρόκειται εδώ για μια ε, μεταρρύθμιση η οποία ε, περιλαμβάνει μέτρα τα οποία απορρέουν από την λιτότητα που έχουν περιπλέξει πάρα πολύ την κατάσταση στην Ιταλία. Σε γενικές γραμμές η μεταρρύθμιση του συστήματος των συντάξεων έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους Ιταλούς πολίτες και επομένως εδώ κατά την άποψή μου έχουμε μία αναφορά η οποία θα πρέπει να μείνει ανοιχτή. Ε, περιμένω βεβαίως και κάποιες επικαιροποιήσεις από την πλευρά της ε, Κομισιόν ε, γιατί πρέπει να, έχει, ε, ε, πρέπει να λάβει υπόψη και την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου της Ιταλίας η οποία έκρινε αντισυνταγματικά ορισμένα τμήματα αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης των συντάξεων. Επομένως θα πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί περιμένοντας τις νέες εξελίξεις. Κάτι άλλο, η κυρία Πιτέρα, παρακαλώ κυρία Πιτέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς θέλουμε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. γιατί δεν ξέρουμε ακόμα με τα βεβαιότητα αν πρόκειται για ε, πρόσκαιρα μέτρα, μεταβατικά ή αν πρόκειται ε, ε, για μόνιμα στοιχεία τα οποία θα σωματωθούν στη μεταρρύθμιση, άρα παραμένει ανοιχτή η αναφορά. Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος, αυτό θα κάνουμε. όλα τα οποια θα σωματωθουν στη μεταρρυθμιση αρα παραμενει ανοιχτη αναφορα πολυ ωραια λεει η προεδρος αυτο θα κανουμε ολα τα θεματα που αφορούν την ισότητα μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και θέλουμε συστηματικά να τα παρακολουθούμε. Αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή εργασία. Πραγματικά σας ευχαριστώ γιατί είχαμε μία δύσκολη μέρα, επιβιώσαμε όλοι. Και αν δεν σας ξαναδώ θα ήθελα να σας ε, πω καλές διακοπές, να σας ευχηθώ καλή ξεκούραση, να μην σκεφτείτε καθόλου την, τις αναφορές και την Επιτροπή, ε, να πιείτε, να φάτε, να διασκεδάσετε, να αλιαστείτε και να περάσετε ωραία.